Bien, mesdames, και κύριοι, καλησπέρα σα Συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή. Ξεκινάμε τη δημόσια ακροασή μα, την οποία διοργανώνει η Υποεπιτροπή μας Ασφάλεια και άμυνα, καθώ επίση και την προσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι σχέσει με το ΝΑΤΟ μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου συνεδριάζουμε, αλλά πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ του 2014, που θα λάβει χώρα λοιπόν το Σεπτέμβριο του 2014 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα μακρηγορήσω. Το ζήτημα το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε καλύψει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα στρατηγικό, το οποίο βλέπουμε σε διάφορα άλλα επιμέρους θέματα ένα ζήτημα το οποίο ανακύπτει συνεχώς. Βλέπουμε ότι ενώ είναι πάρα πολύ απτά τα ζητήματα, προκύπτουν κάποιες δυσκολίες ανυπέρβλητες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να συντονίσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στους δύο αυτούς πυλώνες, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά, γιατί 23 από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν και στο ΝΑΤΟ, διότι ο διάλογος, ο υψηλό είναι ιδιαίτερα έντονος, συχνός, γίνονται πάρα πολλές ε, διασταυρούμενες παρεμβάσεις τόσο του κυρίου Ράσμουσεν όσο και της κυρίας Άστον σε πολλά διαφορετικά φόρα. Έχουμε σαφώς πολλά κοινά συμφέροντα και αναφέρθηκα βέβαια και σαν υπέρεπτες δυσκολίες διότι γνωρίζουμε όλοι τα πολιτικά εμπόδια τα οποία συναντάμε και κυρίως το ότι στις περισσότερες επιχειρήσεις μας καθώς επίσης και στις εργασιακές μας σχέσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια τα οποία παρακολύουν τη συνεργασία μας. Και δυστυχώς δεν μας σε θέση ακόμα να καταρρύψουμε γρήγορα τα εμπόδια αυτά. Οι σχέσεις βέβαια αυτές επηρεάζονται από την γενικότερη βούληση να έχουμε αλληλοσυμπληρώμενες και συντονισμένες δράσεις Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές συμφωνούν ως προς αυτό όσον αφορά την αλληλοσυμπληρωματικότητα, κάτι το οποίο έχουμε πολλές φορές και σε κοινοβουλευτικά μας ψηφίσματα. Απόλυτη αλληλοσυμπληρωματικότητα, ιδέα την οποία προωθούμε πάρα πολύ συχνά και όπου θα κατέληγε ουσιαστικά σε ένα ΝΑΤΟ το οποίο θα ήταν καθαρά στρατιωτικό και μια Ευρωπαϊκή Ένωση καθαρά πολιτική μη στρατιωτική, δεν είναι η καλύτερη δυνατή εκδοχή της συμπληρωματικότητα. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθούμε μια δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα έχει και μια στρατιωτική συνιστόσα. Αν δούμε μάλιστα και τον χάρτη των αποστολών των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αποστολές αυτές περιλαμβάνουν μια στρατιωτική συνιστόσα πέρα από τα όσα μπορεί να κάνει να συμβάλλει το ΝΑΤΟ. Επομένως η έννοια αυτή της συμπληρωματικότητας είναι μια έννοια την οποία θα πρέπει να χειριζόμαστε με αρκετή προσοχή. Ο συντονισμός πάντως, ότι δεν έχει φτάσει τα ανώτερα επίπεδά του σε πολιτικό επίπεδο, γιατί όπως σας είπα υπάρχουν διάφορα εμπόδια και κυρίως ανάμεσα στην Κύπρο και την Τουρκία, παρόλα αυτά περιλαμβάνει μία άλλη συνιστόσα τις στρατιωτικές δυνατότητες, δυνατότητες τις οποίες αποφασίσαμε να καλύψουμε σήμερα με την δημόσια ακρόασή μας. Κατά αυτόν τον τρόμο μπορούμε να συνδυάσουμε περισσότερο αυτά τα οποία γίνονται και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας αλλά και από την ATC του ΝΑΤΟ. Νομίζω λοιπόν ότι η συνεργασία αυτή θα είναι ιδιαίτερα επικοδομητική και θα συμβάλλει και στο pooling and sharing την συνένωση δυνατοτήτων και στην εκμετάλλευση την οποία προωθούμε. Έχουμε δύο τμήματα λοιπόν στην δημόσια κουρασή μας σήμερα το απόγευμα. Το πρώτο πάνελ θα ασχοληθεί με την στρατηγική καθώς επίσης και την ανάπτυξη των ε, στρατιωτικών δυνατοτήτων, ζήτημα το οποίο αποτελεί ε, τμήμα των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τμήμα της ημερήσιας διάταξης της Συνόδου του, ε, του ΝΑΤΟ, ο κύριος Χάινριχ Χιμπράους είναι ο πρώτος ο οποίος θα πάρει το λόγο. Είναι βοηθός γενικός γραμματέας για ζητήματα μεντικού σχεδιασμού και προγραμματισμού στο ΝΑΤΟ λοιπόν. Και έχουμε και τον κύριο Γκος, ο οποίος είναι αναπληρωτής γενικός διευθυντής στον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο πάνελ της ε, δημόσιας ακορασής μας, θα ασχοληθούμε σε αυτό περισσότερο με την έννοια της συμπληρωματικότητα και των συνεργειών που μπορούν να προκύψουν άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Το λόγο θα πάρει ο κύριος Φρό από το ΝΑΤΟ και ο κύριος Ραμπό ο οποίος εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και είναι επικεφαλής της μονάδας ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού στα πλαίσια της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού. Δίνω ευθύ αμέσως το λόγο στον κύριο Μπράους, ο οποίος θα μας μιλήσει για το ζήτημα των δυνατοτήτων. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντονζόν. Ε, φαντάζομαι ότι δεν πειράζει να μιλήσω αγγλικά. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τα ευγενικά σας λόγια με τα οποία με υποδεχθήκατε. Δεν λέω ότι ξαναγυρνάω στα, στο σπίτι μου, αλλά ε, παλιά είχα εργαστεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, επανειλημμένως ερχόμουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ενημέρωση. Τώρα ως εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ ε, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να, να βρίσκομαι εδώ για να, για να μιλήσουμε για τα θέματα που παρουσίασε ήδη ο κύριος Τανζό, δηλαδή για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεργαστούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια παρουσίαση περίπου 10 λεπτών για να σας δώσω την πολιτική μας άποψη σχετικά για τη σχέση ακριβώς Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ στο, ε, σχετικά ακριβώς με το θέμα της ε, ανάπτυξης δυνάμεων και των ε, σχετικών προσπαθειών θα σας δώσω κάποιες πρακτικές συμβουλές μετά για το τι κάναμε μέχρι τώρα και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στο μέλλον. Η άμυνα είναι σημαντική είναι σημαντική και αυτό είπε άλλωστε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Δεκέμβρη. Αυτό για μας είναι πάρα, στο ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι και δική μας πεποίθηση ότι είναι σημαντική η άμυνα. Αυτό το defense matters, δεν ξέρω ποιος έχει το copyright για αυτή τη φράση, αν είναι το Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ τελικά. Λοιπόν, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα ασφάλειας και και αναγνωρίζουμε πλήρως το σημαντικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Ρασμούσεν στο, στο περσινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο φετινό στη φετινή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ε, όπως είπε λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας είναι ότι ε, ε, πρέπει να διαμορφώσουμε μια ισχυρή Ευρώπη η οποία να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ε, προκλήσεις, να είναι δυνατός ε, παίκτη και να μπορεί να σταθεί απέναντι στις Ηνωμένε Πολιτείες. Βεβαίως τον Ιούνιο του 2015 θα πρέπει να ε, κάνουμε αξιολόγηση το κατά πόσον επετέφθησαν οι στόχοι οι οποίοι ετέθησαν. Αυτό θα είναι ένα άλλο ρώσιμο στην ιστορία των σχέσεων των δύο χωρών. Των δύο μερών, με συγχωρείτε. Πέρα λέει όμως από αυτό από αυτά τα γεγονότα τα οποία πραγματικά ε, είναι μεγάλης πολιτικής σημασίας θα πρέπει να ε, καταβάλουμε κοινέ προσπάθειες για να ενισχύσουμε την άμυνα της ε, Ευρώπης το Σεπτέμβρη στην ε, συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και την εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Η... Το ΝΑΤΟ ε, προσβλέπει στο μέλλον. Εδώ και 65 χρόνια έχει ε, αγωνίζεται για τους ίδιους σκοπούς και έχει, και επι, έχει δεχθεί καινούρια μέλη, καινούριους εταίρους τηρώντας βεβαίως και τη στενή επαφή με τους ε, φίλους μας στην απέραντη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε ένα όραμα για το ΝΑΤΟ, θέλουμε ένα ισχυρό ΝΑΤΟ στο μέλλον. Ε, αυτό είναι το ΝΑΤΟ του μέλλοντος για το οποίο μιλάμε και βεβαίως ε, αυτό σχετίζεται με τα, και με τα μέλη μας και με την άλλη πλευρά του ε, Ατλαντικού όπως είπαμε. Στη Λισαβόνα το 2010 στο Σικάγο αργότερα μιλήσαμε για το τι πρέπει να κάνουμε, ορίσαμε το ΝΑΤΟ 2020 ορίσαμε κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορούν οι σύμμαχοι να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν περισσότερο τις δυνάμεις τους και από κοινού αλλά και ο καθένας ξεχωριστά. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις, υπάρχουν κάποια εμπόδια, παρόλα αυτά επιτυγχάνουμε πρόοδο θεωρώ. Ιδιαίτερα για την προοπτική των δυνάμεων το 2020 έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο και η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφή θα εκτιμήσει, θα αποτιμήσει τις προσπάθειες που κάναμε και τα αποτελέσματά τους. Θα... Θέλουμε επίσης και θα ε, να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ότι θα έρθει η ανισορροπία που υπάρχει όσον αφορά την κατανομή των βαρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ευρώπης θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ενισχύσει τις δυνατότητες της και τις δυνάμεις της να ενισχύσει κάνει προσπάθειες ασφάλειας για να προχωρήσει προς την άρση αυτής της ανισομέρειας. Στο... τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ε, σχέση ε, για την πολιτική της Ευρώπης σε θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής ε, ήταν επίσης ένα σημαντικό ορόσημα στην ιστορία. και ε, στις αποφάσεις που πάρθηκαν λέγεται σαφώς ότι χρειάζεται στενότερη συνεργασία μεταξύ ημών και ημών το ε, Αυτά όλα πρέπει να τα λάβετε υπόψη και εσείς αλλά και εμείς προετοιμάζονται στη Σύνοδο Κορυφής του Σεπτεμβρίου. πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις δυνάμεις μας. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα μη επανδρομένα ε, εναέρια οχήματα, τι γίνεται με την εναέρια ανατροφοδότηση. Όλα αυτά είναι θέματα που ξέρουμε σας απασχολούν και εσάς μας απασχολούν και μας. Θα πρέπει να και εσείς και εμείς να τα σκεφτούμε και να, τα, και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα σχετικά μέσα και στις ε, δικές σας αλλά και στις δικές μας ε, επεμβάσεις. Άρα και μακροπρόθεσμα θα πρέπει να φροντίσουμε και η μεν και η δε να προγραμματίζουμε και να σχεδιάζουμε με παρόμοιο τρόπο, με ένα τρόπο συνεκτικό και η smart defense του ΝΑΤΟ και το pooling και sharing της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι συμπληρωματικές πολιτικές. Θα πρέπει να δου, φροντίσουμε να ευθυγραμμίζονται επίσης οι μην άμεσες αντίδραση του ΝΑΤΟ και το battleground της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε παρόμοιες ομάδες, παρόμοιες προσπάθειες κάνουμε και μεν και η ΔΕΕ θα πρέπει να φροντίσουμε να συγκλίνουν οι προσπάθειες αυτές. Η διαδικασία σχεδιασμού του ΝΑΤΟ και η αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστούν περισσότερο και το Νοέμβριο οι Υπουργοί Άμυνας στα συμπεράσματά τους μίλησαν για αυτή την ανάγκη και την ομοιότητα των δύο διαδικασιών που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τους συναδέλφους μας για να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτή η ευθυγράμμιση διότι βεβαίως η διαδικασία λήψη αποφάσεων στους δύο οργανισμούς είναι διακριτή. Θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε τη συνεργασία, να συνεχίσουμε το συντονισμό και αυτό πιστεύουμε ότι θα αποβεί προς όφελος και των δύο. Θα πρέπει να δούμε επίσης το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, την, την προστασία των θαλασσών μας, την ανάπτυξη των δυνάμεών μας. Θα πρέπει να δούμε σε μεγαλύτερο βάθος τι μπορούμε να κάνουμε για τα θέματα αυτά. Σας ανέφερα ήδη αρκετές από τις προτεραιότητες που θεωρεί προτεραιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν μεγάλη σημασία και για μας και ε, στις οποίες πιστεύουμε και εμείς ότι μπορεί να γίνει πρόοδος. Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι πραγματικά με ενθάρρυνε ιδιαίτερα η ετήσια έκθεσή σας για την κοινή πολιτική ασφάλειας και εξωτερικής δράσης 2013 που ε, και ε, αναφέρεται σε μια συμπληρωματική προσέγγιση και στενότερη, ε, στενότερο συντονισμό και αποφυγή επικάλυψη και διπλής δουλειάς. Πιστεύω πραγματικά ότι η ενίσχυση της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ενοχλεί το ΝΑΤΟ και η ανάπτυξη των δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης είναι προς όφελος του ΝΑΤΟ. Εν συντομία θα πρέπει να δράξουμε τις ευκαιρίες που μας δίνουν τα, συμπεράσματα των Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του, της Συνόδου Κορυφής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γκος. Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ κύριε Ντανζό. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω με μια δήλωση του Γενικού Γραμματέου του ΝΑΤΟ του κ. Ράσμοσεν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Είπε λοιπόν ότι αν η Ευρώπη είναι απρόθυμη ή ανίκανη να αναλάβει το ρόλο της στην παγκόσμια σκηνή, κάποιος άλλος θα έρθει και θα καλύψει το κενό της. Επίσης, ο κ. Διπάολο, πρώην Υπουργό Άμυνα ε, τη Ιταλία, περισσότερη Ευρώπη είναι καλή και για το ΝΑΤΟ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αντίπαλος του ΝΑΤΟ, είναι εταίρος. Και έχει τελειώσει πια αυτά τα καλυστία μεταξύ των δύο οργάνων. Και μάλιστα σε περίοδο λιτότητας η επικάλυψη είναι πολυτέλεια για όλους. Άλλωστε τα περισσότερα όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Όπως λοιπόν είπε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο προετοιμάζοντας τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Φυσικά έχουμε κάποια όρια στις δυνατότητές μας εξαιτίας κάποιων πολιτικών εμποδίων που ξεπερνούν την άμυνα. Για παράδειγμα, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα και το ΝΑΤΟ δεν μπορούν επίσημα να συνάψουν συμφωνία. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν και να συνεργαστούν. Φυσικά και μπορούν. Και μάλιστα με ελαστικότητα και ευληγησία μπορούμε να βελτιώσουμε τις την κατάσταση μεταξύ μας προς όφελος όλων των κρατών μελών. Και φυσικά κινητήριο μοχλός είναι ο ρεαλισμός. Θέλουμε να βρούμε λύσεις και να δούμε πώς θα αναπτύξουμε καλύτερα τις ικανότητές μας. Και φυσικά χάρη σε στενές επαφέ με το, μεταξύ του ΝΑΤΟ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα. Για παράδειγμα, ε, ανακάλυψη ταυτότητα. Έχουμε ένα εργαστήριο τέτοιες αποκάλυψης ταυτότητας στο Αφγανιστάν για να έχουμε τεχνικές πληροφορίες ε, από επιθέσεις. Να μπορούσουμε να δούμε ποιες είναι, ποια είναι η διαδικασία παροχής ε, διαβατηρίων ε, στοιχείων ταυτότητας και πιστεύουμε ότι έτσι βοηθήσαμε και, την ISAF. Ελικόπτερα με χάρη στη βοήθεια και του ΕΟΑ Εκπαιδεύσαμε προσωπικό και υπτάμενο ε, προσωπικό για τα ελικόπτερα και πάνω από 250 ε, πιλότοι έκαναν την εκπαίδευση σε εμά και αναπτύχθηκαν μετά στο Αφγανιστάν. Ανεφοδιασμός εν σε καύσιμα. Είμαστε υπέρ ενό πολυεθνικού στόλου δεξαμενό με ισχυρή υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε μόνο 42 τέτοια ε, δεξαμενόπλε στην Ευρώπη και πάνω από 500 στι Ηνωμένε Πολιτείε. Γι' αυτό και εργαζόμαστε στενά και με το ΝΑΤΟ, την αντίστοιχη την οργάνωση του ΝΑΤΟ και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνέργειες στις διάφορες φάσεις του προγράμματος. Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας είμαστε υπέρ των πολυεθνικών ικανοτήτων, διασυμμαχικών και δεν πρόκειται μόνο για τις ικανότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά τις ικανότητες των κρατών μελών που μετά τις δεσμεύουν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κοινέ αποστολές. Και υποστηρίζουμε ε, και δικές μας αποστολές, αλλά και αποστολές του ΝΑΤΟ, όταν υπάρχουν κενά στις ικανότητες. Για παράδειγμα, όπως είπε και ο κύριος Μπράους, το θέμα του εναέριου αναφαντασμιωμένου σε καύσιμα, ε, ε, τηλεπικοινωνίες, ε, επικοινωνίες ε, δορυφορικές και τα λοιπά, τηλεκατευθυνόμενα για παράδειγμα, αεροσκάφη. Θέλουμε να συνεχίσουμε για να έχουμε κοινά στοιχεία που θα έχουν πολλούς στόχους και να, πολλαπλούς στόχους και να εξασφαλίσουν διαλειτουργικότητα. Επίσης, έχουμε κοινή ευθύνη και ε, είμαστε υπόλογοι απέναντι στους φορολογούμενους για το πώς αξιοποιούμε τα κονδύλια, τα, τα κοινοτικά κονδύλια. Βέβαια και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν καλύτερα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Και από αυτή την άποψη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας ε, μπορεί να παράσχει σημαντική βοήθεια. Για παράδειγμα, το θέμα της ε, μεταβλητής γεωμετρίας. Καμία από τις προτάσεις μας και τα σχέδιά μας δεν είναι υποχρεωτικά. Χώρες που επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν και άλλες να αυτοεξαιρεθούν. Έχουμε βέβαια το θέμα της προτυποποίησης και της ε, πιστοποίησης. Αυτά είναι για όλους. Αλλά υπάρχουν και σχέδια που είναι αλακάρτα. Αρκούν δύο χώρες μέλη για να ξεκινήσουν ένα σχέδιο και στη συνέχεια μπορούν να προσχωρήσουν και άλλες. Έτσι υπάρχει ελαστικότητα και καινοτομία. Επίσης, ενημερώνουμε άμεσα τους Υπουργούς Άμυνας ως διακυβερνητική οργάνωση και παρακολουθούμε στενή, στενά τις δραστηριότητες σε υπουργικό επίπεδο και έχουμε ε, και καθοδήγηση αλλά και την ευλογία κατά κάποιο τρόπο του Συμβουλίου Υπουργών. Στην φάση της προετοιμασίας ενός προγράμματος αλλά και στην εκτελεστική φάση έχουμε ε, συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Έτσι μπορούν και τα κράτη-μέλη με πολύ αποτελεσματικό τρόπο να αναπτύσσουν τι ικανότητέ του. Επίση έχουμε στενή σχέση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι που είναι προ όφελο φυσικά και του ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, το θέμα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, ενιαίου ευρωπαϊκή εθέρε. Το ΣΕΖΑΡ θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην άμυνα, σε θέματα άμυνας. Άλλωστε έχουμε και το μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη, πάνω από 2.000 καταδεκτικά, 800 μεταγωγικά και 600 ελικόπτερα. Και μάλιστα το κόστος του Σεζάρ για το το στρατιωτικό κλάδο θα είναι μέχρι και 4 δισεκατομμύρια. Αυτό θα επηρεάσει και το ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, Air Command Control Area, δηλαδή ε, το, το, το πεδίο του, αεροπορικ, του της αεροπορικής, ε, του, του ε, συντορισμού των αεροπορικών επιχειρήσεων. Έτσι πιστεύω θα εξυπηρετήσουμε ταυτόχρονα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό Έχουμε και ένα σχέδιο στρατιωτικής ε, εφαρμογής του ΣΕΖΑΡ με συμμετοχή του Eurocontrol, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Επίσης έχουμε μηχανισμό διαβούλευσης με το ΝΑΤΟ για να έχουμε ενιαίε θέσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε έχουμε εντάξει τον ΝΑΤΟ και σε τακτικό επίπεδο στο ΣΕΖΑΡ και μπορεί να μα κοινοποιήσει τι ανησυχίε του χάρη στον διαμεσολαβητικό ρόλο που είχε ο ΕΟΑ. Και αυτό ε, αποκαλούμε πραγματικά αμοιβαία ενίσχυση. Το θέμα τη εφαρμογή τη οδηγία για, για τι προμήθειε τη άμυνα. Θα είναι σημαντική η επιρροή αυτής της οδηγίας στον ε, στη βιομηχανική βάση και στη συνεργασία στην Ευρώπη. Περιμένω το 2016 τη σχετική έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ήδη συγκεντρώνουμε στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Η οδηγία αυτή θα επηρεάσει και το ΝΑΤΟ. Γιατί στον τομέα αυτό θα μπορούσαμε να είμαστε έντιμοι διαμεσολαβητές μεταξύ τη κοινότητα τη Άμυνα και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες αδυναμίες, κάποια στοιχεία που λείπουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, το, η εντολή που έδωσε το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου να εξεταστούν κάποια κίνητρα για την συνεργασία, αλλά και το θέμα το οικονομικό. Στα τέλη του 2014 θα συντάξουμε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επίσης, αλληλεπίδραση ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την προστιθέμενη αξία. Δεν θα πρέπει να αποσπούν την προσοχή μας συζητήσεις ίσονος σημασία, όπως εναρμόνιση κάποιων σχεδίων προγραμματισμού που είναι κάπως διαφορετικά μεταξύ τους γιατί μπορούμε να συγκλίνουμε, αλλά δεν είναι πανομοιότυπα αυτά τα σχέδιά μας και δεν θα έπρεπε να είναι. Γιατί το ΝΑΤΟ θέλει να έχει στόχους ε, ικανοτήτων για τα μεμονωμένα κράτη. Είναι θέμα εθνικού δηλαδή περισσότερο σχεδιασμού. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστοιχο σχέδιο ανάπτυξη των ικανοτήτων ε, ασχολείται περισσότερο για την ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι συνεργατικό αυτό ο σχεδιασμό και επικεντρώνεται στη διαχείριση των κρίσεων. Φυσικά μπορούμε να εναρμονίσουμε κάποιου μηχανισμού για να συγκεντρώνουμε καλύτερα τι ε, πληροφορίε και να κερδίζουμε και χρόνο. Πέραν τούτο όμω οτιδήποτε θα ήταν ε, υπερβολικό και παρατραβηγμένο. Εν κατακλείδη, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα έχει στενή συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και νομίζω ότι η λέξη κλειδί είναι αποφυγή των επικαλύψεων και συμπληρωματικότητα. Εμείς υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των ικανοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα, το ΝΑΤΟ, ακόμη και τα Ηνωμένα Έθνη. Έχουμε, ενεργούμε και ως γέφυρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΝΑΤΟ και φυσικά θέλουμε στενή συνεργασία εν ώψη προετοιμασίας της επόμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, κυρίως ε, με βάση τα βασικά στοιχεία που θα εξεταστούν εκεί. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να πάρετε το λόγο, Τσάρλς. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω ότι έχω μια πολύ ρεαλιστική προσέγγιση καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής μου καριέρας. Πραγματικά δεν μπορώ να προσεγγίσω τα όσα συζητάμε με τρόπο ιδεολογικό. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να έχουμε τις απαραίτητες στρατιωτικές ικανότητες, ιδίως σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και περιορισμού των αμυντικών προπολογισμών στα περισσότερα κράτη-μέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι όντω ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα συνεργάζεται επικοδομητικά με το ΝΑΤΟ για ζητήματα όπω το pooling and sharing, για την ευφύ άμυνα και το καθεξής. Εφόσον ισχύουν όλα αυτά, τα νέα είναι πολύ θετικά. Ξέρω τα ζητήματα αυτά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα για τη δική μου τη χώρα. Η Βρετανική κυβέρνηση έχει θέσει το ζήτημα της περαιτέρω συμμετοχής και συμβολής στον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε ένα συμπέρασμα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουν ε, συγκεντρωθεί τα απαραίτητα αποδεκτικά στοιχεία ακόμη, προκειμένου να ταχθούμε υπέρ της μίας ή της άλλης λύσης. Πάντως, εφόσον μπορούμε να έχουμε συνεργασία επικοδομητική με τον ΝΑΤΟ, τότε εγώ ως Βρετανός θα ήθελα να υποστηρίξω τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει όντως συμπληρωματικότητα. Και όσο υπάρχει συμπληρωματικότητα, τόσο περισσότεροι Αμερικάνοι θα λένε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη καθώς επίσης και η στάση που έχω σαν αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην, στο ΝΑΤΟ. Χάρηκα πάντως πάρα πολύ που άκουσα τόσο την παρουσίαση του κύριου Μπράους όσο και του κύριου Γκός και προσβλέπω στη συνέχεια της συνεδρίασης αυτής. Σας ευχαριστούμε πολύ Τσάρλς, ο κύριος Πάσκου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις θέλω να θέσω. Πρώτον, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είχε δώσει τέλος σε όλους τους πολέμους και βλέπουμε τώρα ότι βρισκόμαστε σε μια φάση συνεχούς αέναης ειρήνης στην Ευρώπη. Πιστεύετε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Ποια είναι η άποψη του ΝΑΤΟ. Δεν είναι τόσο δεδομένη η ειρήνη αυτή. Δεύτερον, ποια είναι η προσέγγιση του ΝΑΤΟ όσον αφορά την ολοκληρωμένη ελεύθερη Ευρώπη. Έχει επιτευχθεί αυτό. Το στόχο αυτό δεν τον έχουμε ακούσει εδώ και δέκα χρόνια. Είχαμε την κρίση στην Ευρώπη, την, το στρατηγικό επαναπροσανατολισμό στις Ηνωμένε Πολιτείε, και δεν έχουμε ακούσει καθόλου τον αρχικό αυτό στόχο εδώ και δέκα χρόνια. Πρόεδρος, ευχαριστούμε ο Τζέφρι Βαν Όρντεν. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω κάποιους παλιούς φίλους από τον, από τον άτοπο στον ΡΙΚ. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ποια είναι η δική μου η θέση. Πραγματικά εντοπίζω πάρα πολλά προβλήματα στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας καθώς επίσης και όλες τις πολιτικές παρεμβάσεις που έχουμε, που ουσιαστικά έχουν ως στόχο να προωθήσουν στο παγκόσμιο προσκήνιο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πέρα από τη θεωρητική αυτή προσέγγιση να υπάρχει και μια πιο ρεαλιστική πρακτική προσέγγιση για να γίνει η πολιτική αυτή πιο αποδεκτή για τα κράτη-μέλη. Η δική μου κυβέρνηση παραμένει σκεπτική και διστακτική όσον αφορά την πολιτική αυτή και πραγματικά χαίρομαι που βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο αν πραγματικά διαβάστε τα συμπεράσματα, καταλήγουν στο εξή συμπέρασμα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στις μη στρατιωτικές δραστηριότητες και όχι τόσο στις στρατιωτικές. και ουσιαστικά δεν προσυπογράφουν όλους αυτούς τους φιλόδοξους στόχους που είχαμε ακούσει στο παρελθόν πριν τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το pooling and sharing και η ευφύς άμυνα είναι τα ίδια πράγματα ουσιαστικά. Για ποιο λόγο πρέπει ουσιαστικά τα ίδια έθνη, τα ίδια κράτη να έχουν δύο ξεχωριστούς οργανισμούς που κάνουν όμως το ίδιο πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει κατά κάποιο τρόπο να βρει έναν τρόπο να συμβάλλει. Πολλές φορές όμως αυτό είναι εντελώς αυθαίρετο και επιφανειακό. Πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επινοήσει κάποιες εργασίες, κάποια καθήκοντα για να δικαιολογήσει την ύπαρξή της στον στρατιωτικό τομέα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έκανε ούτως ή άλλως το ΝΑΤΟ προτού δημιουργηθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Ξέρετε ότι βέβαια αυτή είναι η φυσιολογική τάση οποιασδήποτε γραφειοκρατία να επεκτείνεται και να δημιουργεί νέα καθήκοντα και νέε αρμοδιότητε. Ωστόσο εγώ δεν είμαι καθόλου πεπισμένο ακόμα για την πολιτική αυτή. Ακόμα και οι εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ πολύ συχνά αναγκάζονται να λένε πόσο χρήσιμη τελικά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ουσιαστικά αυτή τη στάση προωθούν τα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ και αυτό το μήνυμα θέλουν να περάσουν επισήμω προ τα έξω. Αν του μιλήσετε επισήμω όμω το περιθώριο των συνεδριάσεων, έχουν εντελώ διαφορετική άποψη. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη ειλικρίνεια σε όλε αυτέ τι δηλώσει. Μιλάμε για την πρόσφατη ε, επιχείρηση αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία μας. Μην γελιόμαστε, δεν είναι ευρωπαϊκή η αποστολή αυτή, ουσιαστικά γαλλική είναι. Η Γαλλία είχε τη βασική πρωτοβουλία και υπάρχουν κάποιοι σύμμαχοι όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες που συμβάλλουν στον τομέα των μεταφορών. Φαντάζομαι ότι και οι Αμερικάνοι θα συνεισφέρουν με ικανότητες εποπτείας. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να παρουσιάσουμε την επιχείρηση αυτή ως καθαρά ευρωπαϊκή επιχείρηση νομίζω ότι δεν συνεισφέρει σε τίποτα πέρα από, το, πέρα από το να δώσουμε μία λανθασμένη παραπλανητική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, δεν υπάρχει ο απαραίτητο έλεγχος για όλε αυτέ τι αποστολές στι οποίε συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπάμαι πραγματικά, εγώ δεν συμφωνώ με την προσέγγιση που έχετε κύριε Πρόεδρε και νομίζω ότι παραπλανούμε τελικά τον Ευρωπαίο πολίτη, έχουμε πάρα πολλέ επικαλύψει, παταλούμε τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου και ουσιαστικά δεν δίνουμε την πραγματική αληθινή εικόνα των πραγμάτων. Euh, Πρόεδρος, χαιρόμαστε όλοι για τη συνέπεια που βλέπουμε να υπάρχει στις α, παρεμβάσεις του Τζέφρι. Εδώ στιγματίζεται και τη γραφειοκρατία βεβαίω. Δεν ξέρω, πρέπει να το σημειώσουν και οι φίλοι μας από τον ΝΑΤΟ. Η κυρία Κρόνιμπεργκ. Ευχαριστώ. Εγώ θα υιοθετήσω την διαφορετική, εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη από τον κύριο Βανόρντεν. Με αυτά που λέει ο κύριος Βανόρντεν ε, κάνει τελικά τη χώρα μου εικονική χώρα. Ε, η, όταν ε, οι Ηνωμένε Πολιτείες λένε ότι απομακρύνονται από την Ευρώπη. Ε. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Μετά από αυτά που είπε ο Τζέφρι, θα ήθελα να πω και εγώ ορισμένα πράγματα. Μιλάμε επί προσωπικής βάσης και όχι εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας. Να ρωτήσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγαλύτερα, περισσότερα προσόντα και μεγαλύτερα όπλα ένα λεπτό Τζέφρι μη με διακόπτεις λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορισμένα ε, ορισμένα πλεονεκτήματα όχι για τα, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έχει ε, κάνει πολλά πράγματα σε μη στρατιωτικό επίπεδο κλπ. Αυτό σημαίνει ότι ο συνδυασμός αυτών και της κοινή πολιτικής ε, ασφάλειας και άμυνας είναι κάτι παραπάνω από αυτό που έχει και κάνει το ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ πολύ Πρώτα-πρώτα για την αποτελεσματικότητα. Αν μπορούμε να καταδείξουμε ότι υπάρχει συμπληρωματικότητα, εσείς είπατε ότι θα παραμένατε στο στην Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Περί αυτού πρόκειται. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας είναι 10 ετών και πρέπει τελικά να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο και να δείξει ότι κάνει κάτι επιπλέον, προσφέρει μια προστιθέμενη αξία. Κύριε Βαντεν Όρντεν, εγώ βεβαίως έχω διαφορετική άποψη από τη δική σας, ούτως ή άλλως διαφωνούμε στην προσέγγιση μας. Εγώ πιστεύω στην συμπληρωματικότητα, δεν πιστεύω στην επικάλυψη ή τη διπλή δουλειά που δεν χρειάζεται. Αλλά υπάρχουν άλλοι τομεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει άλλα πράγματα από ό,τι κάνει το ΝΑΤΟ. Παραδείγματο χάρη στι μεταφορέ. Ε, κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Τώρα όμω μα ζητήθηκε από ότι Μα είπαν οι Ηνωμένε Πολιτείε, φροντίστε να καλύψετε ήδη τι ανάγκε σα. Εμείς πια απομακρυνόμαστε. Άρα υπάρχει ανάγκη η Ευρώπη να σηκώσει το γάντι, να ανταποκριθεί στην πρόκληση και να κάνει κάτι πιο συγκεκριμένο. Είπα για το Σεζάρ παραδείγματος χάριν ότι ε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και πραγματικά το ΝΑΤΟ αν συμμετάσχει στην κοινή αυτή η κοινοπραξία σε θα έχει να προσφέρει κάποια πράγματα. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε άλλα και ίσως και παραπάνω. Το μόνο στο οποίο μπορώ να, όπου μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας ήταν ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ουσιαστικά ήταν ε, μια πολιτική εφεύρεση, εφεύρεση για πολιτικούς λόγους. Ωραία, αλλά ακόμη και αν ήταν εφεύρεση για πολιτικούς λόγους αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταυρώσουμε τα χέρια. Έχει ε, πρόκειται για ένα οργανισμό με 120-125 άτομα ε, προσωπικό και 30 εκατομμύρια προπολογισμό. Δεν μπορείτε να μας συγκρίνετε με τον ΝΑΤΟ. Δεν θέλουμε να συγκριθούμε με τον ΝΑΤΟ. Αν βεβαίως προσπαθούσαμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο όσον αφορά το σχεδιασμό με αυτό που κάνει το ΝΑΤΟ θα αποτυχάναμε δεν θα κάναμε σωστή δουλειά εμείς ε, ε, είμαστε άλλου είδους οργανισμός από ότι είναι το ΝΑΤΟ συμπληρωματικότητα λοιπόν και κυρία Κρόνμπεργκ λέτε ότι απομακρύνεται η, η, απομακρύνονται οι Ηνωμένε Πολιτείε από την Ευρώπη. Πώς επηρεάζει αυτό τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Και ναι και όχι. Διπλωματική απάντηση θα μου πείτε. Αλλά εμείς πραγματικά θέλουμε να συνεχίσουμε εκείνα και τα προγράμματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να καλύψουμε τις ανάγκες εκείνες που είναι πραγματικές και που δεν καλύπτουν πλέον οι Ηνωμένε Πολιτείε, όπως παραδείγματος χάνει ένα αέρια ανατροφοδότηση που είπε το ΝΑΤΟ. Ο κύριος Μπράουζερ τώρα έχει το λόγο. Σίγουρα. Δεν αισθάνομαι σε θέση να προσπίσω εγώ την ε, κοινή, την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Το 2014, 100 χρόνια μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρισκόμαστε ιστορική σίγουρα επέτειος και φυσικά και ταυτόχρονα ορόσημο στην πορεία του ΝΑΤΟ προς το 2020 και την ε, μεταρρύθμισή του προκειμένου να δημιουργηθεί ε, μια δέσμη δυνάμεων που θα είναι διαλειτουργική, ε, πολλαπλών καθηκόντων που θα μπορεί να αναπτυχθεί παντού υπό κάθε περίσταση και σε συνεργασία με τους εταίρους. Αυτό είναι ο στόχος μας ε, κατά τη μεταρρύθμιση του ΝΑΤΟ. Και τώρα γνωρίζουμε ότι ε, σίγουρα η ειρήνη είναι ένα πολύτιμο αγαθό και θα πρέπει οπωσδήποτε να την ε, διαφυλάξουμε στην Ευρώπη. Είμαι Γερμανός και ο Χέλμοντ Κόλ, πρώην καγκελάριος, ε, πίστευε και εγώ το πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να, διαφυλάξουν, ε, θέλει να διαφυλάξει την ειρήνη στην Ευρώπη και από κοινού με το ΝΑΤΟ θέλουμε να διαφυλάξουμε την ειρήνη και στην Ευρώπη και για την Ευρώπη. Και πιστεύω στο στόχο αυτό. Και κατά τη γνώμη μου το ΝΑΤΟ έχει τρεις βασικές αποστολές. Συλλογική άμυνα, διαχείριση των κρίσεων και ε, ασφάλεια που στηρίζεται στη συνεργασία. Και σίγουρα η συλλογική ασφάλεια και η άμυνα είναι σημαντικό θέμα, παρόλο που δεν είναι προφανές, είναι βάση και ακρογωνίως λίθος του γενεσιουργού λόγου, του λόγου ύπαρξης ουσιαστικά του ΝΑΤΟ. Δεν συμφωνώ απόλυτα εδώ με τον συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν εστιαζόμαστε μόνο σε συλλογικές ε, επιχειρήσεις ασφάλειας. Δεν έχουμε ε, ειδικέ ικανότητε για συλλογική άμυνα και όλα τα άλλα είναι για τη διαχείριση των κρίσεων. Όλα είναι περίπου για το ίδιο. Και θα πρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη. Είτε στην περιφέρεια του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης, για παράδειγμα Τουρκία. Εκεί είχαμε την ανάπτυξη συστημάτων Patriot ε, στα σύνορα από τρεις ε, συμμάχους του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα δύο από αυτές τις χώρες ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ανταποκρινόμαστε λοιπόν σε περιστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Και φυσικά έχουμε και το θέμα της ε, ειρήνης και της ασφάλειας μάλλον εκτός της Ευρώπης που μπορεί όμως να επηρεάσει την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία εντός της Ευρώπης. Η Ευρώπη ε, που θα είναι ελεύθερη Χόουλεντ κέρι και Ελεύθερη του Πατρός Μπούς. Πολύ σημαντικό θέμα. Και το θέμα είναι να αφήσουμε ανοιχτές τις πόρτες μας ε, ε, και στη, όχι μόνο προς τα μέλη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και προς τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και θα παραμείνουν ανοιχτές οι πύλες μας και θα δείτε ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία θα κάνει σαφείς δηλώσεις και θα δώσει και υποσχέσεις Τούτου λεχθέντος έχουμε δύο γύρους διευρύνσεων που τις έχουμε ξεπεράσει. Τώρα έχουμε 28 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και έχουμε σαφείς παραμέτρους και αρχές και συγκριτικούς κανόνες, benchmark, με βάση τους οποίους θα αξιολογήσουμε οποιαδήποτε περαιτέρω υποψηφιότητα και αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Γιατί θα πρέπει σίγουρα και πρώτα απ' όλα να βελτιώσουμε τη συλλογική μας άμυνα. Οπότε μια χώρα θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε θέση να συμβάλλει στη σταθερότητα, την ειρήνη και την ελευθερία στην περιοχή της. Και αν έχουμε υπόψη και την Ευρώπη αλλά και την ευρύτερη περιοχή, όλα αυτά τα θέματα δεν είναι εύκολα να τα αναλάβει μόνη της οποιαδήποτε χώρα. Γι' αυτό και ίσως είναι εύλογη η επιθυμία εισαγωγής ε, ένταξης στο ΝΑΤΟ. Οπότε Σίγουρα κάθε περίπτωση θα εξεταστεί ενδελεχώς και μεμονωμένα. Δεν υπάρχουν καθόλου προϋποθέσεις. Και αν παρακολουθήσετε και τα ανακοινωθέντα τύπου και τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέως μας, η, η αρχή είναι ότι κάθε χώρα είναι ελεύθερη και έχει απόλυτη ελευθερία επιλογής ε, ε, και δυνατότητα να διαλέξει τους συμμάχους της. Αυτό είναι δεδομένο. Και στην πράξη αναζητούμε συμφωνία μεταξύ 28 χωρών όταν κάποιος ε, χτυπάει την πόρτα μας και θέλει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. CSDP, Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Θα έλεγα ότι εγώ είμαι υπάλληλο ε, διοικητικό ε, με ορολογία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με ορολογία του ΝΑΤΟ, θα έλεγα ότι είμαι μέλο του διεθνού προσωπικού. Υπηρετώ το αφεντικό μου. Το αφεντικό μου είναι 28 χώρε μέλη ουσιαστικά. Και θα συμφωνείτε ότι στο πλαίσιο αυτό Απορρίπτω οποιοδήποτε υπενιγμό ότι δηλώσεις οποιοδήποτε ε, από τις 28 χώρες ε, ε, για, την, για την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα ότι είναι ανέντιμη δεν θα μπορούσα να δεχτώ οποιαδήποτε τέτοια νήξη υπενιγμό. Μια και το ΝΑΤΟ είναι η συμμαχία 28 χωρών στην οποία συμμετέχει και το Ηνωμένο Βασίλειο και στη διακήρυξη του Σικάγο φαίνεται ότι η κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα και προσπάθεια προσπάθειε Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, για την κοινή μα ασφάλεια, είναι πολύ σημαντική συμβολή στην κοινή μα ασφάλεια. Εγώ πιστεύω ακράδαντα σε αυτό, σε αυτή τη διακήρυξη και είναι σαφή δήλωση που σε καμία περίπτωση θα πρέπει να την ε, υποτιμούμε, να την απαξιώνουμε ακόμη και οι Αμερικανοί στο ΝΑΤΟ, δήλωσαν με σαφήνεια ότι δεν ενδιαφέρονται όπου, πότε και με ποιο τρόπο οι Ευρωπαίοι θα αναπτύξουν πραγματικές σημαντικές ικανότητες. Το πιο σημαντικό είναι να το κάνουν και όχι με ποιο τρόπο και πού και πότε. Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Και ως προς την ερώτηση της προστιθέμενης αξίας της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. η βασική της προστιθέμενη αξία είναι αυτή η σφαιρική, η ολιστική προσέγγιση. Τουλάχιστον στη θεωρία. Έχουμε ένα τεράστιο φάσμα εργαλείων και ε, ιδεών που μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στη διαχείριση των κρίσεων. Και το ΝΑΤΟ ε, έχει ως βασική δύναμη το στρατιωτικό σκέλος. Και το βασικό χαρακτηριστικό είναι η διάρθρωση το, της αλυσίδας ε, ε Και θα πρέπει να είμαστε σε θέση συνεχώς ε, να σχεδιάζουμε για τα πάντα και να δίνουμε στους πολιτικούς ηγέτες πολύ γρήγορα ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών προκειμένου να σχεδιάσουμε και να ολοκληρώσουμε απαιτητικέ και μεγάλε ευέλικτε επιχειρήσει. Αυτό κάνει το ΝΑΤΟ και αυτό δεν δίνεται να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αυτή, αυτό το σθένο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δύναμη τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια προσέγγιση που είναι πολιτικο-στρατιωτική και όχι μόνο στρατιωτική όπω είναι του ΝΑΤΟ. Και είναι μοναδική αυτή η ιδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα και εμεί υπολογίζουμε σε αυτήν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένε χώρε και περιοχέ που το ΝΑΤΟ για πολλούς και διάφορους λόγους δεν έχει. Για παράδειγμα Γεωργία. Πολλές χώρες στην Αφρική. Αυτό μπορεί να αλλάξει το μέλλον, αλλά προς το παρόν το ΝΑΤΟ δεν έχει ουσιαστική πρόσβαση σε όλες αυτές τις περιοχές. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναπτύξει πολύ αποτελεσματικά μέσα, αστυνο, αστυνομικές δυνάμεις, ε, εμπειρογνώμονες για το κράτος δικαίου. Είναι τεράστιο το δυναμικό που έχει εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΝΑΤΟ το αναγνωρίζει αυτό το δυναμικό. Επίσης έχουμε ολοκληρώσει ε, και μία ιδέα της δικής μας σφαιρικής προσέγγισης που αξιοποιεί το δικό μας στένος, τη δική μας δύναμη και την προθυμία και τιμότητά μας για στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα Ηνωμένα Έθνη και μάλιστα για συνεργασία επιτόπου. Και αν το κάνουμε με αποτελεσματικό τρόπο αν συνεργαστούμε με αποτελεσματικό τρόπο, τα αποτελέσματα θα είναι πραγματικά απαράμιλα και ως προς τα θέματα της διαχείρισης των κρίσεων και της πρόληψης των, κρίσεων. Θα επανέλθουμε στο θέμα των ικανότητων. Πάντως σίγουρα πιστεύουμε στην προστιθέμενη αξία της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Και όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ την έχουν αναγνωρίσει και την έχουν αξιοποιήσει. Είναι δεδομένη αυτή η προστιθέμενη αξία και η συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε... Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ζέλερ θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας βρίσκεται μέσα στις συνθήκες μας και ε, ακόμη και δεν το πιστεύουν ορισμένοι συνάδελφοι λίγο λίγο θα γίνει πραγματικότητα ε, υπήρχε ο ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, το τείχος του Βερολίνου που δεν υπάρχει πια ε, και προσπάθεια τότε που έγινε να ε, προστατεύσουμε τον ε, δυτικό κόσμο από το τις δυνάμεις της Ανατολής που απειλούσαν με μια έννοια τη Δυτική Ευρώπη οι Αμερικάνοι βοήθησαν τώρα έχουν αρχίσει να απομακρύνονται όλα αυτά συνέβησαν ωστόσο αγαπητοί συνάδελφοι ο κόσμος μας δεν έγινε πιο ειρηνικός πιστεύουμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση λίγο λίγο κουράζεται όλο και περισσότερο επειδή καλείται να επιλύσει αντιπαραθέσεις και σειράξεις στη, έξω από, το εσωτερικό της αν θέλετε και, και ε, ε, ξέρετε πολύ καλά ορισμένα πράγματα που έγιναν πρόσφατα, τις ικανότητες στρατιωτικές των ευρωπαϊκών δυνάμεων που τελικά ξεκίνησαν οι Γάλλοι με ορισμένα αεροπλάνα και μετά ε, αναγκαστήκαμε να ρίξουμε βόμβες και αυτό απέδειξε ότι τελικά η, Ευρωπα... η Ευρώπη δεν ήταν αρκετά ικανή όσο νόμιζε. Ναι, θα πρέπει λοιπόν να τα συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά και να δούμε ότι απαιτείται στενή συνεργασία. Ε, με το ΝΑΤΟ για την προστασία της υπήρου μας. Από την άλλη μεριά βεβαίως έχουμε επιχειρήσεις που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία παραδείγματος χάρη και γίνεται η προσπάθεια να καλυφθούν ε, κάποιες ε, ε, δαπάνες από τα ε, κονδύλια ε, ανάπτυξη και συνεργασία στην ανάπτυξη. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να βελτιωθούν και να αλλάξουν. Και η θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να καθίσουν να σκεφτούν πιθανές λύσεις και μαζί με, μαζί με το ΝΑΤΟ, μαζί με τις ΗΠΑ να αναζητήσουν τις λύσεις αλλά κατά κύριο λόγο να φροντίσουν να ενισχύσουν τις δικές τους δυνάμεις. Πέρασαν οι εποχές της απεικιοκρατίας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ορισμένα πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε. Εκείνα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε τουλάχιστον να τα κάνουμε από κοινού σε συνεργασία η χώρα μου, η Γερμανία, αναγνώρισε επιτέλους ότι τέλειωσε η μεταπολιτική περίοδος και για μας και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε συνεργασία με άλλους. Ευχαριστούμε κύριο Σκόβα. Ευχαριστώ. Δεν είχα την πρόθεση να λάβω το λόγο, αλλά μου κίνησε το ενδιαφέρον το παράδειγμα που δώσετε με τη Γεωργία και τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Διάβασα το κείμενο του Ράσμουσεν που λέει ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να φτάσει μέχρι τον Κάφκος από πολιτική άποψη. Και ίσως εκεί θα ήταν ένα καλό πεδίο συνεργασίας. Γιατί έχουμε ήδη προχωρημένες διαπραγματεύσεις πολιτικές το θέμα της συμφωνίας σύνδεσης και μάλιστα η κοινή γνώμη της Γεωργίας είναι υπέρ της ένταξης του ΝΑΤΟ, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για στενή συνεργασία της χώρας αυτής ε, με το ΝΑΤΟ. Βέβαια, έχουμε και την Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου, αλλά έχουμε συγκεκριμένη κατάσταση. Ο γείτονα της ε, Γεωργίας ε, είναι πολύ κοντά σε 11 χιλιόμετρα, οπότε... Δεν ξέρω αν μπορούμε μαζί με τον ΝΑΤΟ να κάνουμε κάτι, γιατί η φήμη μας στην Γεωργία, η φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γεωργία είναι δεν είναι και πολύ καλή. Δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, γιατί δυστυχώς η Γεωργία θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να επηρεάσει την κατάσταση ώστε ο βόρειος ε, γείτονας της ε, ε, Γεωργίας να μην θέσει τα σύνορα εκεί που ήθελε. Οπότε αυτή την άποψη δεν χαίρομαι ιδιαίτερη εκτίμηση στην κοινή γνώμη της Γεωργίας. Βέβαια, σε κάτι τέτοιο ακόμη και ο κύριος Βανόρ θα μπορούσε να συνενέσει. Τι θα μπορούσαμε εμείς πραγματικά να κάνουμε εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το παράδειγμα που δώσατε με τη Γεωργία. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι μπορούμε να σας δώσουμε μια ομόφωνη συγκεκριμένη απάντηση από το ΝΑΤΟ όσον αφορά τη Γεωργία αναφέρομαι τουλάχιστον στην απάντηση που θα μπορούσε να σας δώσει το ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω πραγματικά ποια δράση θα μπορούσε να λάβει το ΝΑΤΟ πέρα από τον να κηρύξει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Ξέρετε το ΝΑΤΟ δεν είναι πολιτική οργάνωση, είναι στρατιωτική οργάνωση. Νομίζω ότι α, αυτό ουσιαστικά σας λέγαμε στην απάντηση την οποία σας δώσαμε πριν από λίγο το ΝΑΤΟ επικεντρώνεται κυρίω εκεί πέρα που υπάρχει στρατιωτική δέσμευση. Ένα λεπτό. Φυσικά δεν μίλησα για στρατιωτική επέμβαση. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μόνο δύο επιλογέ, στρατιωτική επέμβαση ή σιωπή. Έχουμε δυνατότητα και πολιτική επιρροή. Άλλωστε, έχουμε συνεργασία με τη Ρωσία, οπότε θα μπορούσαμε και εδώ μιλούμε και για συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Θα μπορούσαμε εκεί από κοινού να ασκήσουμε την αποτελεσματική μας ε, επιρροή. Γιατί εκεί υπάρχει μεγαλύτερο φάσμα επιλογών σε ό,τι αφορά την πολιτική επιρροή. Και νομίζω ότι πραγματικά κατάφορα παραβιάζονται όλοι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου μπροστά στα μάτια μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να αρκούμαστε στο γεγονός ότι α, επειδή διαλέγουμε τη στρατιωτική επέμβαση η μόνη άλλη εναλλακτική που έχουμε είναι η σιωπή. Όχι, υπάρχει και άλλη λύση πέραν της στρατιωτικής επέμβασης. Ε, συγγνώμη, σας είπα ότι οι διεθνείς οργανισμοί έχουν συγκεκριμένε εντολές. Το ΝΑΤΟ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ασκεί πολιτική πίεση σε μια χώρα. Διαφορετικά καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ψηφίσουν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ για να αλλάξει η αρμοδιότητα του οργανισμού αυτού και πραγματικά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ δεν πρόκειται ομόφωνα να συμφωνήσουν ποτέ για κάτι τέτοιο. Κάθε διεθνής οργανισμός έχει την εντολή του και τις συγκεκριμένες αρμοδιότητές του. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Ο κύριος Μπράους. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς έχουν ως κοινό στόχο την σταθεροποίηση, τη διατήρηση της ειρήνης και αυτό ισχύει και για την Ευρώπη. Εσείς αναφερθήκατε κυρίως τώρα στην άποψη που υποστηρίζουν οι Αμερικάνοι. Ξέρετε τι είχε πει ο Ρόμπερτ Γκέιτς, όχι ο Μπιλ Γκέιτς, διορθώνει ο μιλήτης. Το 2011 ο πρώην Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ είχε πει ότι Ευρωπαίοι πραγματικά πρέπει να κάνετε περισσότερα πράγματα για τη δική σας την ασφάλεια. Εμείς εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες είπε δεν είμαστε πλέον σε θέση να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα όποτε εσείς μας χρειάζεστε για τη δική σας τη διατήρηση ασφάλειας και είπε επίση ότι ανησυχούσε για το γεγονός ότι είχε δημιουργηθεί μια συμμαχία δύο διαφορετικών κατηγοριών. Από τη μια οι Ηνωμένε Πολιτείε και από την άλλη πλευρά όλες οι υπόλοιπε ε, χώρες. Ξέρετε ότι ε, ορισμένοι άλλοι θύνοντες είχαν πει ότι υπάρχουν κάποιοι καλοί στρατοί αλλά με μέγεθος μπονζάι, πολύ μικρό στην Ευρώπη. Αν λοιπόν εξετάσετε την κατάσταση ορισμένων χωρών είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στο ΝΑΤΟ, στην Ευρώπη βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες που έχουν πλέον στρατούς που πειράζονται πάρα πολύ από την έντονη οικονομική κρίση που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό αποτελεί πολύ μεγάλη πρόκληση. Και δεν σας το λέω όλα αυτά για να επιτύχουμε αυτή την καλύτερη δυνατή εξισορρόπηση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Κάνω τις δηλώσεις αυτές γιατί πιστεύω ότι και η ίδια η Ευρώπη θα πρέπει να αποτελεί έναν αξιόλογο εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η σχέση αυτή η συνεργασία αυτή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικέ προκλήσεις. Αλλά από την άλλη η Ευρώπη θα πρέπει να είναι σε θέση και μόνη της να λαμβάνει δράση όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Να φερθήκατε στην κρίση στη Λιβύη. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να είχαμε διεξάγει την επιχείρηση αυτή με τον τρόπο που το κάναμε, δηλαδή τόσο αποτελεσματικά και τόσο σύντομα, τόσο γρήγορα, αν δεν μας είχαν υποστηρίξει στα παρασκήνια ουσιαστικά οι Ηνωμένε Πολιτείε, δίνοντάς μας απαραίτητες στρατιωτικές ικανότητες. Και στη συνέχεια αυτό το οποίο μας είπανε εσείς Ευρωπαίοι που συμμετέχετε στο ΝΑΤΟ να ξέρετε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Πρέπει να είστε σε θέση από μόνοι σας να αναλάβετε δράση. Ενδεχομένως να προκύψουν περιπτώσεις στο μέλλον όπου οι Ευρωπαίοι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα πλαίσια του ΝΑΤΟ θα πρέπει να αναλάβουν δράση από μόνοι τους. Έχοντας βέβαια μια κάποια υποστήριξη από τους Αμερικάνους, αλλά όχι τόσο ισχυρή υποστήριξη όσο στο παρελθόν. Νομίζω ότι και αυτή την αλλαγή ισορροπίας πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η ευρωπαϊκή οι Ευρωπαίοι, με συγχωρείτε, σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, είτε ενεργούν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, είτε ενεργούν στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορούν να κάνουν από μόνο του περισσότερα πράγματα. Το πλεονέκτημα λοιπόν του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα είναι ότι είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να έχει μεγαλύτερη επιρροή ή μεγαλύτερη διασύνδεση, αν θέλετε, τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία. Επομένως, αποτελεί σημείο επαφής και για μας σε υπηρεσιακό επίπεδο από πλευράς ΝΑΤΟ για να καταφέρουμε να συνεργαζόμαστε καλύτερα με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να πετυχαίνουμε καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τις ικανότητες των Ευρωπαίων είτε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ όσον αφορά τώρα τη Γεωργία. Chatham House εδώ πέρα είναι μια δημόσια ακρόαση, επομένω πρέπει να είμαι πιο διπλωματικός. Όταν είπα πρόσβαση του ΝΑΤΟ στην Γεωργία, αναφερόμουν στο 2008, μετά τον πόλεμο δηλαδή στη Γεωργία. Εκείνη λοιπόν την εποχή, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πρόσβαση στην ουσία. Πρέπει ωστόσο να πω ότι η Γεωργία είναι ένας πολύτιμος αξιόλογος εταίρος του ΝΑΤΟ η συμβολή τους στις επιχειρήσεις μας θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι εντυπωσιακή θα έλεγα. Όποτε μπορούν συμβάλλουν στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Όποτε μπορούν με τις δικές τους τις δυνατότητες προσπαθούν να ενδυναμώσουν τις σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Γεωργίας με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και αυτό όντως έχει αναγνωριστεί από το ΝΑΤΟ, έχει εκτιμηθεί από το ΝΑΤΟ και εμεί θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις εταιρικέ αυτές σχέσεις που έχουμε με τη Γεωργία. Τώρα, στη χώρα αυτή, άνω του 70, 75% από όσο γνωρίζω των ανθρώπων των πολιτών είναι υπέρ του ΝΑΤΟ. Δεν θα έλεγα ότι είναι μοναδικό αυτό, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός σε σχέση με άλλες χώρες και αναφέρομαι και σε κάποιους παραδοσιακούς ε, συμμάχους ε, του ΝΑΤΟ, παραδοσιακά μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή και κλεισμένο των θυρών στο ΝΑΤΟ θέλουμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με την Γεωργία αλλά και με άλλες χώρες εταίρους. Και ελπίζουμε, ή ελπίζουν στη Γεωργία, ότι κάποια στιγμή, όχι στο τόσο μακρινό μέλλον, θα τους δοθεί η δυνατότητα να αρχίσουν να συζητούν και την ενδεχόμενη προσχώρησή του στο ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνετε ότι από πολιτική πλευρά το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Είμαστε σε πολύ στενή σχέση με τι αρχέ τη Γεωργία. Πρέπει πάντω να σα πω ότι η Γεωργία είναι ένα ιδιαίτερα αναγνωρισμένο εταίρο πλέον του ΝΑΤΟ και δεν έχει ένα πολιτικό απλώς διάλογο με το ΝΑΤΟ, αλλά όπως σας είπα συμβάλλει σε καθημερινή βάση στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και στις συζητήσεις που διεξάγονται στο ΝΑΤΟ. Και ξέρετε ότι υπάρχει και μία στρατηγική, σύμφωνα με την οποία ενισχύοντας τις εταιρικές μας σχέσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός Ευρώπης, είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε την πολιτική μας για τη σταθερότητα, για την παγίωση και την εδραίωση της σταθερότητας, από το να επεμβαίνουμε τοπικά σε κάποιες περιοχές. Θεωρούμε ότι προϊόντος του χρόνου πετυχαίνουμε πολύ περισσότερα πράγματα συνάπτοντας εταιρικέ σχέσεις και όχι επεμβαίνοντας αναγκαστικά στρατιωτικά. Δύο ακόμη παρεμβάσεις. Λαντμπέργκης και Όρντεν και μετά κλείνουμε το πρώτο αυτό πάνελ. Κύριε Λαντμπέργκης και μετά θα αναλάβει την Προεδρία ο κ. Παλέτσκι, ο αντιπρόεδρός μας. Λαντσμπέργκη. Αν το ΝΑΤΟ είναι υπέρ της ειρήνης, αυτό δεν είναι πολιτική θέση. Γιατί δεν είναι πολιτικός στόχος το να έχουμε ειρήνη και να αγωνιζόμαστε για την ειρήνη μπορούμε να πάμε και παρακάτω το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να εφαρμόζει να επιβάλλει πολιτική πίεση Μα ε, είναι πόλεμος. Ο πόλεμος τι είναι, είναι πολιτική δράση και μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος χωρίς ε, ε, πίεση. Θέλω να πω ότι αυτά τα σλόγγαν είναι λίγο μη πραγματικά. Τώρα για τις αμυντικές ικανότητες του ΝΑΤΟ, είτε γίνεται διεύρυνση είτε όχι. Εγώ προέρχομαι από τη Λιθουανία τα αντίστοιχα θέματα α, αντιμετωπίζαμε και πριν από πολλά χρόνια. Μπορούμε, είμαστε ικανοί να υπεραμεινθούμε το εαυτού μας ή όχι. Ή Τώρα για τις αρχές, πολιτικές, ηθικές και άλλες αυτές είναι δεδομένες αλλά αυτή η ε, ικανότητα άμυνας πέρα από αυτές τις αρχές χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σαν κριτήριο για να γίνει μια χώρα μέλος ή όχι και η ετοιμότητα αναφέρεται σε ετοιμότητα του ΝΑΤΟ. Ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να αναλάβει το κίνδυνο ή το βάρος να ε, προστατεύσει μια χώρα. θα μπορούσαμε να καταλάβουμε βέβαια αν αυτή η ε, προσέγγιση του ΝΑΤΟ ήταν ε, σήμαινε λιγότερα θα μπορούσε να δικαιολογηθεί λέει το ΝΑΤΟ όσο λιγότερα μέλη τόσο λιγότερα προβλήματα εντάξει αλλά το λέει το ΝΑΤΟ αυτό Είπατε παρακάτω ότι η γεωργία είναι πολύ κάνω καλός συνεισφορέας σε τι στις ανάγκες μας. Ωραία. Και βάζετε τελεία εκεί. Εκείνοι τι, τι ανάγκες έχουν. Θέλουν ειρήνη οι άνθρωποι. Αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ας τους να συνεισφέρουν και εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Φοβάμαι ότι το ΝΑΤΟ, ότι σε έναν κόσμο όπου οι, οι δημοκρατίες δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητές στις μη δημοκρατίες το ΝΑΤΟ τι κάνει προσπαθεί να παρεμποδίσει κάποιους γείτονες ε, οι οποίοι έχουν επεκτατικές τάσεις. Εγώ θυμάμαι παλιά, παλιά το ΝΑΤΟ ε, ήθελε να διασφαλίσει ασφάλεια, να προστατεύσει τις χώρες κτλ. Μετά ο Γέλτσιν είπε πάρτε την Πολωνία αλλά όχι τις βαλτικές χώρες. Και ο Κλίντον είπε όχι. Ήταν πολύ σημαντική η χρονική στιγμή αυτή. Σήμερα όμως, τι γίνεται στο Βουκουρέστι για τη Γεωργία οι Ηνωμένε Πολιτείε παρέμειναν στις ίδιες βασικές γραμμές. Η ε, Ευρώπη άλλαξε στάση. Και τι έγινε. διότι μιλάμε για αμυντικές ικανότητες αλλά οι ικανότητες η άμυνα δεν σχετίζεται μόνο σε ηλικιές δεν έχει μόνο ηλική υπόσταση έχει και μια πνευματική διάσταση είμαστε έτοιμοι θέλουμε πιστεύουμε ότι μπορούμε να ε, προστατεύσουμε κάποιον να βοηθήσουμε ή παραμυνθούμε κάποιου το ΝΑΤΟ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έχει κατά νου το ΝΑΤΟ ε, ε, πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαστεί τι είναι ποιος δεν ε, Πρέπει οπωσδήποτε να διατηρήσουμε την πνευματική πτυχή αυτή του θέματος. Βαν Όρντεν, πρόεδρε, συμφωνώ ότι οι Αμερικανοί είπαν δεν μας ενδιαφέρει πως το οργανωθούν οι Ευρωπαίοι φτάνει να έχουν παραπάνω ικανότητες και να τις χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες αυτές ε, για την άμυνά τους η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρώπη λάβετε υπόψη σας η Ευρωπαϊκή Ήπειρος εσείς σαν ΝΑΤΟ πείτε μας τι θα ζητούσατε από μια άλλη αν θέλετε οργάνωση αντίστοιχη με τη δική σας που, που μπορεί να τη λέγανε Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα ζητάγατε εγώ τι θα έλεγα θα έλεγα πραγματική συμπληρωματικότητα, ισότιμη κατανομή καθηκόντων εργασιών υποχρεώσεων, η συνεργασία στην ανάπτυξη μετά την οποιαδήποτε ενόπλη σύραξη παραδείγματος χάρη μετά από οποιαδήποτε καταστροφή κοινό προγραμματισμό στο μέλλον Δεν θέλουμε, αυτό θέλουμε, να θα έπρεπε να πει το ΝΑΤΟ. Δεν θέλουμε να έχουμε δύο παράλληλες δομές και εκπρόσωπους ε, στη Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην αντίστοιχη του ΝΑΤΟ ε, ε, που να ζουν κάποια αντιπαλότητα φαντάζομαι, ανταγωνισμό μεταξύ τους. Κύριε Φανόρντεν, Ίσως ε, το αποτέλεσμα θα σας εξέπλητε αν είχα μια εξουσιοδότηση εν λευκό. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι η ερώτηση είναι μάλλον ουτοπική και πολύ τεχνητή, ρητορική σχεδόν. Το ΝΑΤΟ το... ιδρύθηκε το 1949. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με και η κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα με τη σημερινή τη μορφή πολύ αργότερα. Ω υπάλληλο όμω του ΝΑΤΟ, οφείλω να αναγνωρίσω ότι τα μέλη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 28 ε, χώρες μέλη, συνυπόγραψαν την ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Και αν δείτε ε, Στη συνθήκη τη Λισαβόνα βλέπετε ότι πολλέ διατάξει δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη, αλλά οι φιλοδοξίε ήταν υψηλέ και πολύ καλά συγκροτημένες και διατυπωμένε. Και αυτό μπορώ, δεν μπορώ παρά να το αναγνωρίσω και να το λάβω υπόψη. Και ω αξιωματούχο του ΝΑΤΟ θα έλεγα ότι αν δούμε καρπούς αυτές τις προσπάθειες, πλεονεκτήματα, συμπληρωματικότητα και προστιθέμενη αξία, τι άλλο θέλουμε, τόσο το καλύτερο και δεν αμφισβητώ το πολιτικό πλαίσιο. Αν καταφέραμε στην Ευρώπη να κάνουμε τις υποψηφιότητες και τη συμμετοχή συνεπή, γιατί έχουμε, έχουμε την Νορβηγία στο ΝΑΤΟ, ενώ δεν είναι η Νορβηγία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε και την Τουρκία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και επίσης δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το αντίστροφο, έχουμε την Κύπρο που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μάλτα, η Ιρλανδία, η Αυστρία, η Σουηδία, η Φιλανδία. Επίσης δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Αλλά είναι κυρίαρχα κράτη και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την πραγματικότητα θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Σουηδία, Φιλανδία, Αυστρία είναι πολύ σημαντική και προσιλωμένη εταίροι στο ΝΑΤΟ, για να αναφέρω μόνο μερικά παραδείγματα. Και φυσικά αποκομίζουμε πολλά ωφέλη από τη συνεργασία αυτή. Αναγνωρίζουμε όμως ότι πολιτικός πώς ε, οι δύο οργανώσεις είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Και ο τρόπος με τον οποίο παρέχουν και εξασφαλίζουν την ασφάλεια είναι κάπως διαφορετικός. Και οι φιλοδοξίε είναι κάπως διαφορετικέ. Θα πρέπει όμω να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη συνεργασία. Και ένα προσωπικό σχόλιο. Δεν βοηθά, κατά τη γνώμη μου, να συνεχίζουμε να μεμψημυρούμε ε, ή να έχουμε μόνο παράπονα για τι εξελίξει. Εγώ λέω καλύτερα να αξιοποιήσουμε την κατάσταση στο έπακρο, στη συνεργασία με τους συναδέλφους της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Γιατί η Ευρωπαϊκή Άμυνα είναι προς το συμφέρον και του ΝΑΤΟ. Και θέλουμε να ενισχύσουμε και τη διατλαντική εταιρική σχέση. Και τον διατλαντικό δεσμό. Κύριε Λαντσμπέργκης, κάνατε κάποιες παρατηρήσεις και θέσατε και απορίες, ερωτήσεις. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα από πολλούς άλλους πόσο δύσκολο είναι το θέμα και πόσο πολιτικά ευαίσθητο. Και είναι εντός του πλαισίου του ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ δεν είναι μόνο αμυντικός οργανισμός. Είναι πολιτικό στρατιωτικός οργανισμός. Και θα είδατε στο παρελθόν τις στεναρές δηλώσεις του Γενικού Γραμματέως για την κατάσταση στη Γεωργία από το 2008 και μετά. Εμείς συνεχίζουμε να επισημαίνουμε αυτό το θέμα στη Ρωσία στα, στις στα κοινά συμβούλια για την κατάσταση στη Γεωργία και την προκαλούμε τη Ρωσία. Γνωρίζουμε την κατάσταση, γνωρίζουμε τις δηλώσεις και μερικές φορές είναι ε, πολύ διαφορετική διάγνωση της κατάστασης και συμφωνούμε ότι διαφωνούμε απλώς μερικές φορές. Αλλά αυτό γίνεται και στο Συμβούλιο ε, ΝΑΤΟ-Ρωσίας και κλεισμένων των θυρών, αλλά πολύ συχνά ήταν κατηγορηματικός ο Γενικός Γραμματέας της ε, δημόσιας δηλώσεις του για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα το μέλλον της Γεωργίας, σε σχέση με το ΝΑΤΟ, η Γεωργία είναι μία από τις τέσσερις χώρες που, έχει, που έχουν βλέψεις να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτές οι τέσσερις χώρες διαφέρουν μεταξύ τους και βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές. Η πολιτική τους κατάσταση και η εγχώρια κατάσταση είναι διαφορετική. Η στρατιωτική τους συνεισφορά επίσης είναι διαφορετική. Η αμυντική τους θεσμή είναι διαφορετική. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις βάλουμε σε δύο τσουβάλι ουσιαστικά, να τις χειριστούμε από κοινού και να ε, ζητήσουμε από τις 28 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ το πράσινο φως για την υποψηφιότητά τους. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και 26 ευρωπαϊκές χώρες που θα πρέπει να καταλήξουν στην ίδια στρατηγική αξιολόγηση με εσά. Αλλά οι απόψεις διαφέρουν και εγώ ως υπάλληλο του ΝΑΤΟ θα πρέπει να το λάβω υπόψη αυτό. Και σας διαβεβαιώ ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ προσπαθεί να θέσει το θέμα στη συζητήση με τις 28 χώρες με ανοιχτό, δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο. Και υπάρχουν πολλοί υποστηρικτέ ε, της γεωργίας στο ΝΑΤΟ. Δημοσίως δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπράους. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο δεύτερο τμήμα της ε, ακροασής μας, στο δεύτερο πάνελ με μια κάποια καθυστέρηση θα, ζητήσουμε, θα συζητήσουμε ζητήματα συμπληρωματικότητα και συνεργειών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ όσον αφορά την συνεργασία σε διάφορες επιχειρήσεις, σε διάφορα θέατρα επιχειρήσεων. Η καταπολέμηση, για παράδειγμα, της πειρατείας στον Ινδικό ωκεανό. Έχουμε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις, την Ocean Shield του ΝΑΤΟ και την EU Αταλάντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο αυτές επιχειρήσεις ε, μπορούμε να πούμε ότι έχουν εστευθεί με επιτυχία, αλλά πώς οριοθετούν ακριβώς τα καθήκοντα και αρμοδιότητες, πώς μπορούμε να μεταφράσουμε τη συνέργεια αυτή και τη συμπληρωματικότητα σε έμπρακτη ε, συμβολή σε διάφορες άλλες επιχειρήσεις που θα έχουμε στο μέλλον. Ο κύριος ε, Φρόχ, Ρίτσαρτ Φρόχ από το ΝΑΤΟ είναι αναπληρωτής βοηθός γενικός γραμματέας αρμόδιος για ζητήματα επιχειρήσεων και του δίνω αυτής αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πέρασα 15-17 χρόνια της επαγγελματικής μου ζωής στο ΝΑΤΟ, ασχολούμενος με ζητήματα ικανοτήτων. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα λοιπόν το πρώτο τμήμα της δημόσιας ακροασής σας και από το 2011 και μετά είμαι πλέον αξιωματικός αρμόδιος για ζητήματα επιχειρήσεων στο ΝΑΤΟ. Βλέπω λοιπόν πραγματικά που ενεργοποιούμεθα ως οργανισμοί. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά στοιχεία που δικαιολογούν τελικά τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ όσον αφορά τις ε, ικανότητες και όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, πάρα πολλές δηλώσεις που αναφέρονται σε αυτή την διατλαντική συνεργασία. Πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουμε έναν πολυδιάστατο, πολυσονοριακό, διασυνοριακό, με συγχωρείτε, κόσμο που υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ κρίσει που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μονομένα από ένα κράτο μέλο. Ουδέποτε μάλλον συνέβαινε κάτι τέτοιο. Απαιτούνται πλέον συντονισμένε συλλογικέ προσπάθειε. Νομίζω ότι ακόμα και οι Ηνωμένε Πολιτείε συνειδητοποιούν πλέον ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνε του. Θεωρούμε πάντως ότι οι συλλογικές αυτές επιχειρήσεις θα πρέπει να ενισχύονται από τις απαραίτητες στρατιωτικές ικανότητες. Αν δεν υπάρχουν ικανότητες αυτές, τότε δεν μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και τίθεται να αμφιβόλω η αξιοπιστία τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ. Κάθε φορά που από κοινού προσπαθούν να διεξάγουν μεγάλες επιχειρήσεις. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των ικανοτήτων, των νέων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, αλλά δεν, δεν αναφέρονται σχεδόν καθόλου στις επιχειρήσεις. Δεν, δεν θα πρέπει να έχουμε ικανότητες μόνο και μόνο για να επικερδίσει αμυντική βιομηχανία, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητες για να καταφέρουμε τελικά να αποτρέψουμε τις κρίσεις και αν προκύψουν οι κρίσεις να τις αντιμετωπίσουμε στρατιωτικά. Ακριβώς επ' αυτού η συνεργασία των δύο οργανώσεων μας είναι πάρα πολύ πλούσια και έχουμε ανταλλαγές σε πάρα πολλά επίπεδα. Είπα ότι εκπρόσωπος και γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, στο δικό μου επίπεδο των βοηθών αναπληρωτών γενικών γραμματέων συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά μαζί με τον Διευθυντή από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Μεντικού Σχεδιασμού ασχολούμεθα με διάφορα θέατρα επιχειρήσεων και έχουν ενταθεί οι συζητήσεις μας για περαιτέρω συνεργασία. Συντοποιούμε ότι εποφελούμεθα και οι δύο από την κοινή αυτή συνεργασία. Στις Βρυξέλλες αλλά και στο ΝΑΤΟ συνειδητοποιούμε ότι στα πλαίσια των θεάτρων επιχειρήσεων αυτών μπορεί πραγματικά να αποβεί η επικοδομητική συνεργασία μας. Τέτοια συνεργασία είχαμε στο Αφγανιστάν, έχει στεφθεί με επιτυχία. Σε θεσμικό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αναθεωρούν το ρόλο τους για την περίοδο μετά το 2014. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις εθνικές ε, αρχές του Αφγανιστάν με μια υποστήριξη περισσότερο για το στρατό της χώρας αυτής στην αποστολή μετά το 2014 θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να καταρτήσουμε την αστυνομία της χώρας στο υψηλότερο επίπεδο προκειμένου να καταφέρουν να αναπτύσσονται επιχειρησιακά σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να καταστήσουμε την αστυνομία της χώρας αυτής από μια αστυνομία η οποία ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη και αναπτυσσόταν σε συγκεκριμένα μέρη της χώρας σε μια πραγματική αστυνομική δύναμη μεγάλου βεληνικούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να επιτελούμε τις αρμοδιότητές μας στα πλαίσια του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών 1244 και το ΝΟΑΤΟ θα συνεχίσει επίσης να συμβάλλει και σε άλλες επιχειρήσεις όπως το Κωσυφοπαίδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και από πολιτικής πλευράς όμως μια σύγκληση και όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμβολή της ύπα της εκπροσώπου έχει διδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η κοινή αποστολή K4ULEX στο Κωσυφοπαίδιο έχει σημειώσει πάρα πολλές επιτυχίες. Έχουμε εκεί ένα πολύ ε, μια πολύ στενή συνεργασία, πολύ καλές επικοινωνίες, καθώς επίσης και πάρα πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στους δύο διοικητές. Μαζί με τον ΟΑΣΑ και τα Ηνωμένα Έθνη καταβάλουμε πολύ σημαντικές διεθνείς προσπάθειες στο Κωσυφοπαίδιο. Ξέρετε ότι ε, πάντα θα υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θα αντιτίθενται στη δική μας την προσπάθεια στην περιοχή αυτή. Πιστεύουμε πάντως όμως με τον επικοδομητικό διάλογο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ καθώς επίσης και με την προσέγγιση που υπάρχει πλέον μεταξύ Πριστίνας και Βελιγραδίου τα πράγματα θα εξελιχθούν θετικά. Η αναθεώρηση τώρα της αποστολής αυτής που θα έρθει σύντομα, καθώς επίσης και οι εκλογές στην περιοχή αυτή θα περάσουν τη μελλοντική εξέλιξη των πραγμάτων. Να μιλήσουμε τώρα για την πολιτική ασφάλεια στη θάλασσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, με την ηγετική δύναμη των ΗΠΑ αναπτύσσονται σε διάφορες περιοχές, ιδίως στα νυχτά της Σομαλίας, προκειμένου να καταπολεμήσουν ε, την πειρατεία. Αναφέρομαι σε συλλογική δράση, γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που συμμετέχουν. Πάρα πολλοί μας καταγγέλουν ότι είναι ότι υπάρχει πληθώρα τελικά παραγόντων και ότι ενδεχομένω να γινόμαστε κάπω αντιπαραγωγικοί. Αλλά τελικά ακριβώ το αντίθετο βλέπουμε στην πράξη. Βλέπουμε ότι πολύ συχνά ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα απαραίτητα πολεμικά πλοία, έρχεται το ΝΑΤΟ να συμπληρώσει. Όταν το ΝΑΤΟ υπολείπεται σε κάποιε στρατιωτικέ ικανότητε, μπορεί να επαφείεται στη συμβολή και τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιώντας τώρα στο Μπαχρέιν την αποστολή μας ΣΕΙΔ έχουμε και εκεί πολύ θετικά αποτελέσματα. Στο μέλλον θέλουμε να επεκτείνουμε για δύο ακόμα χρόνια μέχρι το 2016 την αποστολή Αταλάντα. Συζητάμε επίσης το μέλλον της αποστολής μας Ocean Shield πέρα από το 2014. Υπάρχει ένα συλλογικό συμφέρον τόσο για τον ΝΑΤΟ όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχιστεί αυτή η εξαιρετική συνεργασία και το ΝΑΤΟ χαιρετίζει τον πολύ καλό ρόλο που είχε αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Σομαλία, στην οικοδόμηση ικανοτήτων και χαιρετίζουμε επίσης και την γενικότερη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της πειρατείας, η οποία θα συνεχιστεί και το 2014 στα νυχτά της Σομαλίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα μεταξύ των δύο οργανισμών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίω σήμερα, γιατί οι πόροι μας μειώνονται όλο και περισσότερο και στις δύο πλευρές, αντικατοπτρίζοντας την οικονομική πραγματικότητα. Πρέπει εμεί να βοηθήσουμε μεν τους δε, προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε τους στόχους μας. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ να έχουν μια κοινή προσέγγιση. Αν συμβεί αυτό τότε όλη η διεθνή κοινότητα μπορεί να αποφεληθεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φρό. Και θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μπερνάρ Ραμπό, ο οποίος είναι επικεφαλής του ε, ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω πράγματα που ελέγχθησαν, να είμαι συμπληρωματικός. Θα σας πω το πολύ συγκεκριμένα τι γίνεται με τη συνεργασία με στα πλαίσια της διαχείρισης ε, <clears throat> κρίσεων ε, πώς προχωρούμε. Αυτή η συνεργασία πρώτα πρώτα να πω ότι πάει καλά και θα περιγράψω λιγάκι το παράδειγμα της Σομαλίας και της καταπολέμης της πειραστίας. Ξέρετε ότι εκεί υπάρχει, ε, υπάρχουν δύο επιχειρήσεις, Ocean Shield και Talante. Από το 2008 υπάρχει μια πραγματικά μοναδική συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο επιχειρήσεων. Ε? Περιλαμβάνονται Εκεί όμως και τη, ο ε, θαλάσσιος αν θέλετε ε, και οι άλλοι φορείς που ασχολούνται με τη θάλασσα και τους θα, θαλάσσιους πόρους ε, εμείς αναλάβαμε την Προεδρία μετά αναλαμβάνουμε τώρα την Προεδρία μετά από την προ, τους Αμερικανούς και ε, Πραγματικά πρέπει να το λάβετε αυτό υπόψη για να καταλάβετε τη συνεργασία ανοιχτά της Σομαλίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Τώρα, να πω επίσης ότι για να προστατεύσει και να περιπολίσει κανείς σε μια ζώνη σαν και αυτή χρειάζεται κόσμο και σκάφη στη θάλασσα τρία-τέσσερα σκάφη μόνιμα έχει το ΝΑΤΟ εκεί. Τα 5 με 8 έχει η, επιχείρηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχείρηση Αταλάντη. Αυτά δεν αρκούν. Πρέπει να προσθέσουμε εκεί και τα αμερικάνικα σκάφη και τα κινέζικα και τα ρώσικα και τελικά έχουμε γύρω στα 30 σκάφη στην περιοχή αυτή. Ε? Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δρούν σε εκείνη την περιοχή. Αυτό θα ήταν ε, μη τίμιο εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν όλοι συνεισφέρουν και όλοι ελπίζουν ότι θα επωφεληθούν και η Ocean Shield και η Atalant ε, είναι σημαντικές πολύ ως επιχειρήσεις από εκεί και πέρα η ύπαρξη της μιας δεν αφαιρεί τίποτε από τη σημασία της άλλης και ε, υπάρχει πολύ στενή συνεργασία και μεταξύ των ηγετών μας, των γραμματέων μας, της ΥΠΑ, του εκπροσώπου κλπ. κλπ όλοι προσπαθούμε να βοηθήσουμε για να υποφεληθούμε με τον καλύτερο τρόπο. Για την Αταλάντη να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα ή στις 28 του μηνός, δεν θυμάμαι ακριβώς, ε, προγραμματίζεται λοιπόν για το την επιχείρηση Αταλάντη η επόμενη συνάντηση. Ε. Γίνεται πολύ σε τακτά χρονικά διαστήματα και πολύ συχνά μια τέτοια συνάντηση. Από εκεί και πέρα υπάρχει το γενικό επιτελείο του ΝΑΤΟ Μαρκόμ ε, και η συνεργασία είναι καθημερινή. Ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών, δεδομένων διαχέονται λοιπόν διαδίδονται όλα τα στοιχεία αυτά προς όλη τη διεθνή κοινότητα ε, άλλο επίπεδο τώρα συνεργασίας είναι, για την προστασία της θάλασσας είναι το εξής. Ε, Προσπαθούμε να έχουμε μια κοινή εποπτική εικόνα της περιοχής και αυτό διευκολύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την επιχείρηση Αταλάντ, αλλά και από τους Κινέζους και άλλους, όπου μέσω ε, υπάρχει σχετικά ε, το κέντρο συλλογής πληροφοριών στο κέρας της Αφρικής και μέσω αυτού του κέντρου διαχέονται, συλλέγονται και διαχέονται και διαδίδονται οι πληροφορίες και τα δεδομένα αυτά. Ε, και από εκεί και πέρα η. Προεδρία ε, ε, αναλαμβάνεται εκ περιτροπής από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται προγραμματισμός ανά δύο-τρεις μήνες. Λοιπόν, αυτή είναι η δομή, θα σας πω τώρα ακριβώ τι γίνεται και θα ήθελα να κρίνετε εσείς μόνοι σας ε, πώς λειτουργούν τα πράγματα. Δεν χρειάζεται νομίζω να προσθέσω τίποτα, τα πράγματα πάνε καλά. Εμείς ουσιαστικά βεβαίως συνεχίζει την πειρατεία αλλά σπάσαμε αν θέλετε το business model που υπάρχει εκεί και ελπίζουμε πολύ γρήγορα να ε, ε να κάνουμε ε, να, και άλλα πράγματα. Τώρα, Πέδιο, Λιβύη, Αφγανιστάν, θα μπορούσα να σας πω χίλια δύο πράγματα για τις επιχειρήσεις εκεί, αλλά θα ήταν υπερβολικά. Ε, συνεργαζόμαστε και σε επιτελικό επίπεδο και σε επίπεδο σχεδιασμού και προγραμματισμού και επί του πεδίου, πρακτικά. Η σχέση μας είναι σχέση εμπιστοσύνης και από εκεί και πέρα στο Κωσιβό πεδίο ε, φτάσαμε στο σημείο να οργανώσουμε ε, το Νοέμβριο και Δεκέμβριο τις ε, ε τοπικές και περιφερειακές εκλογές άρα υπάρχει στενή συνεργασία. Τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πήρε κάποιες αποφάσεις όπως είπαμε το Δεκέμβριο του 2012. Υπάρχουν χίλια δυο πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά και σίγουρα η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι οργανώσεις μας είναι ε, τεράστιες. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, από εκεί και πέρα ποιος έχει κάποια πλεονεκτήματα σε ποια σημεία ε, γιατί υπάρχουν κάποιες διαφορές. Από την άλλη μεριά όμως πραγματικά γίνεται η συνεργασία είναι καλή και ε, εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα στην Αφρική ασχολούμεθα ιδιαίτερα και στηρίζοντας κάποιες επιχειρησιακές δράσεις αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης κτλ. και με στα πλαίσια της ε, ομάδας ε, ε, ταχείας αντίδρασης. Σας ευχαριστώ. What about questions Θα ακούσουμε λοιπόν τις ερωτήσεις προς τους δύο καλεσμένους μας και φαντάζομαι ότι είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να απαντήσουν. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι καλές Αναφερθήκατε στην επιχείρηση Αταλάντη για τη Σομαλία. Θυμάμαι όμως σχετικά μια παλιότερη συνεδρίαση όπου ο επικεφαλής της Αταλάντα ήρθε εδώ και μας είπε ότι η καταπολέμηση της πειρατείας θα πρέπει να συνδυαστεί με το γεγονός ότι μεγάλα σκάφη ευρωπαϊκών χωρών ε, βρίσκονται στην περιοχή και υπεραλλιεύουν. Αν, θα αν μπορούσαν να συνδυαστούν λοιπόν, η ε, να συνδυαστούν η καταπολέμηση της πειρατείας με αυτή της υπεραλίας αυτό θα ήταν προς το συμφέρον των πολιτών των χωρών που, για τις εκτές των οποίων μιλάμε. Ε, είναι γεγονός βεβαίως ότι κάποιες ε, ε, ακτές αφρικανικές ε, γίνονται αντικείμενο υπερεκμετάλλευση και υπεραλίας αυτό μπορούμε να το αμφισβητήσουμε και εκεί φταίνε οι Ευρωπαίοι Εν πάση περιπτώσει αυτό σε παρένθεση είπα απλώς τι λέει ο επικεφαλής Αταλάντε. Τώρα πιστεύω λοιπόν ότι η συνεργασία αυτή να το Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική και νο, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να διευρυνθεί η συνεργασία αυτή να μην πρόκειται μόνο για στρατοικές δράσεις αλλά και για ανθρωπιστική βοήθεια για κοινωνική στήριξη και για κοινωνικές σχέσεις νομίζω ότι κάτι τέτοια, κάποιες τέτοιες δράσεις αξίζει να αναλυφθούν δεν ε, μπορούμε να αναλαμβάνουμε κάποιες πρωτοβουλίες και να γνωρούμε κάποιες άλλες οι οποίες όμως υπάρχουν και είναι προς το καλό των πολιτών. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς παρακαλώ. Κυρία Νέτς. Ευχαριστώ. Ακούγοντάς σας, Καταλάβουμε ότι γενικώ ε, επιτόπου τουλάχιστον υπάρχουν πολύ καλές ε, σχέσεις μεταξύ των δύο εταίρων. Βέβαια, έχουμε πολύ διαφορετικές ε, περιστάσεις στο Κωσυφοπαίδιο και στο Πακιστάν και έτσι και παρά τις διαφορές επιτόπου η συνεργασία συνεχίζεται. Τώρα για, το όρο ΣΥΝΑ ε, και το Σαχέλ. Βρίσκονται αυτές οι δύο περιοχές στο πολιτικό σα ραντάρ. Γιατί ε, διαβάσαμε την έκθεση της Human Rights Watch για φρικαλαιότητες που καθημερινά λαμβάνουν χώρα στο όρο Σινά, όπου οργανωμένες συμμορίες πάγουν ε, υποψήφιους πρόσφυγες από την Ερυθρέα που προσπαθούν να περάσουν μέσα από τη Σομαλία και να φτάσουν στις όχθες της Μεσογείου και φυσικά αυτό το θέμα διακυβεύει την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Ε, Διαρωτώ με λοιπόν αν ε, σας απασχολεί καθόλου αυτή η κατάσταση, αν θα μεριμνήσετε ενδεχομένω αν θα επέμβετε στις δύο περιοχές, στο Σεχέλ και στο Ρωσινά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση. Ακούγοντα τι ομιλίε σα, διαπιστώνουμε ότι η συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής, Επιτροπής, ε, και Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ΕΔΑ είναι ιδεώδης. Είχαμε τις δύο επιχειρήσεις της Αταλάντης εκ μέρου Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του Ocean Shield της ασπίδα του ωκεανού εκ μέρου του ΝΑΤΟ. Εκεί συμμετείχαν και Ρώσοι και Κινέζοι. Παρ' όλα αυτά εκεί υπήρξαν κάποιε παρεξηγήσει και μας μιλήσατε για κάποια στρατιωτικά μυστικά. Μπορείτε όμως παρόλα αυτά να μας πείτε ποιες ήταν οι δυσκολίες αυτής της ε, επιχείρησης και πού εκεί δημιουργήθηκαν προβλήματα, χωρίς να παραβιάζετε φυσικά στρατιωτικά μυστικά. Τώρα, τι γίνεται με το σχεδιασμό νέων αποστολών. Για παράδειγμα, στον κόλπο της Γουινέας υπάρχουν κάποιες ε, προθέσεις για τέτοια μελλοντική συνεργασία στα σημεία αυτά. Καταρχήν, <laughs> αισθάνομαι σαν να πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη που πάνε τόσο καλά οι σχέσεις μεταξύ μας, γιατί σίγουρα οι χαρμόσυνες ειδήσεις δεν πουλάνε εφημερίδες, αλλά <laughs> τι να σας πω, μπορώ να σας απογοητεύω, πάντως οι σχέσεις μεταξύ μας είναι πολύ καλές. Δεν ήταν ανέκαθεν έτσι και στη... Ένα τμήμα της τετρονίας μας ασχοληθήκαμε τις ικανότητες και συμμετείχα σε πολλές συνεδριάσεις της αρμόδιας ομάδας και εκεί όντως αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, δυσκολίες συντονισμού. Αλλά στις επιχειρήσεις έχουμε κοινούς στόχους για την καταπολέμηση της πειρατείας. Έχουμε τόση πολλή δουλειά που μπορούμε κάλλιστα να την καταμερίσουμε μεταξύ μας και υπάρχει τεράστια ανάγκη συντονισμού. Ξεκινήσαμε πολύ δραστήριο και έντονο συντονισμό για το κοσυφοπαίδιο κατά την έναρξη του διαλόγου Πρίστινας Βελιγραδίου. Και ο, η κυρία η, ο κύριος Ράσμουσεν και ο υπέξ του, της, των Ηνωμένων Πολιτειών μας είπαν πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και προσπαθήσαμε μετά από εντολή να δούμε τι γίνεται ακριβώ και να εξασφαλίσουμε το μέγιστο δυνατό συντονισμό μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικέ ε, φορέ χρειάστηκε να ε, συναντιόμαστε κάθε 15 μέρε. Τώρα έχει επιβραδυνθεί αυτή η συχνότητα των επαφών. Αλλά είχαμε ανέκαθεν ε, σε τακτικό επίπεδο πολύ καλούς δεσμούς. Στις Βρυξέλλες είχαμε πολλές επαφές και αυτή, αυτό το επίπεδο συντονισμού λειτουργεί θαυμάσια. Τώρα, εδώ και τρία χρόνια ασχολούμαι με την καταπολέμηση της πειρατείας και ήμουν στην ε, ομάδα εργασίας ε, για την ε, καταπολέμηση πειρατείας στις όχθες της Σομαλίας, στις ακτές Σομαλίας και μερικές φορές στο, ε, λόγος της πειρατείας ήταν η υπεραλήψη ή η απόρριψη τοξικών αποβλήτων. Αυτό εξωθεί μερικές φορές τους νέους της Σομαλίας να μπαίνουν στη θάλασσα και να ασχολούνται με την πειρατεία. Μπορεί να αληθεύει κάτι τέτοιο, μπορεί και όχι. Μπορεί να υπάρχει πάντω έστω και ένα μικρό τμήμα αλήθεια. Γιατί όντω η πειρατεία είναι επικερδή δραστηριότητα. Εγκληματική μεν, αξιόπινη. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή την ανάλυση κάποιο ίχνος αλήθεια πρέπει να υπάρχει. Και το θέμα τη υπεραλήψη. Θα πρέπει αυτά να το δούμε Όλα από εκείνο γιατί η δημόσια κοινότητα βρέθηκε εκεί ε, κυρίως ε, λόγω της αλίας γιατί εξαιτίας της πειρατείας ε, δισεκατομμύρια δολάρια χάνονται γιατί χρειάζεται να πάνω από όλο δρόμο τα πλοία να καταβάλουν ενισχυμένα ασφάλιστρα και για όλα αυτά φυσικά επιβαρύνονται οι καταναλωτές σε τελική ανάλυση. Ήταν μεγάλο το οικονομικό διακύβευμα, γι' αυτό και έσπευσε η διεθνής κοινότητα εκεί. Βέβαια, πολλέ φορέ όταν έχουμε προβλήματα στη θάλασσα, οι λύσεις τους ε, βρίσκονται στην ξηρά. Γι' αυτό και κάτι πρέπει να κάνουμε. Και έχουμε το, ένα συγκεκριμένο σχέδιο, Νέστορ, και ήμουν την περασμένη εβδομάδα σχετικές συνομιλίες και ένα από τα θέματα ήταν η Σομαλία και η καταπολέμηση της πειρατείας. Όλες οι διεθνείς ε, οργανώσεις και οργανισμοί πρέπει να συμμετέχουν και να κάνουν ό,τι μπορούν. Ο καθένας από την πλευρά του και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πολλά κοινά σημεία. Έχουν και διαφορές βέβαια. Ακούσαμε τον κύριο Μπράους ε, που είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια ισχυρά σημεία που δεν τα έχει το ΝΑΤΟ, ενώ το ΝΑΤΟ έχει αντίστοιχα ισχυρά σημεία που δεν τα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να να αλληλοβοηθηθούμε. δεν ξέρω αν μιλήσατε για το... Εσείς μιλήσατε για το Πακιστάν, εγώ είπα, ανέφερα ως παράδειγμα το Αφγανιστάν. Για τις Αιχέλες ή μάλλον την περιοχή του Σαχέλ, έχουμε ευθύνη για, πολιτική, για στρατηγική παρακολούθηση των εξελίξεων στον κόσμο, αλλά κυρίως ε, στην Ευρώπη και την περιφέρεια της Ευρώπης. Οπότε η Σαχέλ ως ζώνη, ως περιοχή μας ενδιαφέρει. Και στον Μεσογειακό Διάλογο έχουμε εταίρους από χώρες της Αφρικής και οι σύμμαχοί μας που βρίσκονται στην νότια όχθη της, στην, ε, στις όχθες Μεσογείου αναγνωρίζουν ότι η Βόρεια Αφρική είναι σημαντική πηγή αστάθειας. Οπότε εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική μπορεί να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη Νότια Ευρώπη και ταυτόχρονα μετά να επεκταθούν στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Οπότε, ναι δεν σχεδιάζουμε επιχειρήσεις εκεί, αλλά παρακολουθούμε σίγουρα την κατάσταση. Και αν αποφασίσουν οι χώρες μέλη να εξετάσουν το θέμα για πιθανή επιχείρηση, θα πρέπει να κινητοποιηθεί όλη η διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την επιχείρηση ασπίδα του ωκεανού, Ocean Shield, στα τέλη του περασμένου έτους έρχεσαμε να έχουμε εταίρους. Μέχρι τότε οι σύμμαχοι ε, μας έδιναν πλοία για την επιχείρηση αυτή. Πέρυσι είχαμε και εταιρική σχέση με την Ουκρανία, έστειλε και αυτή η πλοία. Ούτω ή άλλως με την Ουκρανία έχουμε και επιχείρηση στη Μεσόγειο κατά πολέμηση τρομοκρατίας που ξεκίνησε το 2001. Active Endeavor λέγεται αυτή η επιχείρηση. Συμμετείχαν ε, και οι Ρώσοι. Τώρα έχουμε ε, την Ocean Shield, την ασφίδα των ωκεανού και μάλιστα και η, η Νέα Ζηλανδία έστειλε ε, πλοίο. Οι Ρουμάνοι, οι Ινδοί, οι Πακιστανοί, όλοι βρίσκονται εκεί, δίνουν το παρόν. Έχουμε τέσσερις ομάδες ε, πολεμικού ναυτικού που βρίσκονται στα... στις όχθες της Σομαλίας. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε ε, την Ocean Shield του ΝΑΤΟ, μια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών και του independent deployers, τι ανεξάρτητε δυνάμει, όπω η Ιαπωνία που από μόνες τους έρχονται και στο Τζιμπουτί επισκέφθηκα ένα Ιαπωνέζικο απόσπασμα. Η πρώτη ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων της Ιαπωνίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταπληκτική οργάνωση, ε, τεράστιος επαγγελματισμός, έχουν δύο πλοία και δύο ε, αεροπλάνα συνέχεια εκεί, τρία ελικόπτερα είναι ανεξάρτητοι όμως, δεν εντάσσονται σε, κανένα, σε καμία άλλη επιχείρηση. Και προσπαθούμε τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε συντονισμό μεταξύ όλων αυτών των φορέων και των κρατών και έχουμε τέσσερα πραγματικά διαφορετικά αποσπάσματα πολεμικού ε, ναυτικού. Και πραγματικά από τις 12 Μαΐου 2012 δεν είχαμε καμία ε, επιτυχημένη απόπειρα πειρατείας. Τις εξουδετερώσαμε όλες και έχουμε επίσης και αποτελεσματικό μηχανισμό αστυνόμευση. και έτσι όταν γίνονται οι απόπειρες εμείς βρισκόμαστε εκεί και τις αναχαιτίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Ραμπό. Κοιτάξτε, τα περισσότερα πράγματα τα έχουμε ήδη καλύψει. Όσον αφορά την καταπολέμηση της πειρατείας μέσω της επιχείρησης Αταλάντα, είναι μια επιχείρηση η οποία ασχολείται και με όλα τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει όσον αφορά την υπεραλίευση, τα οποία στη συνέχεια υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει μια άλλη δραστηριότητα στην οποία δεν αναφέρθηκα στα πλαίσια αυτής της ολιστικής προσέγγισης για την περιοχή αυτή. Έχουμε και την αποστολή UCAP στο κέρας Αφρικής όπου προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις θαλάσσιες ικανότητες των χωρών αυτών μέσω περιπολίας ε, για την ε, εξασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των χωρών αυτών Βλέπουμε ότι ε, από το 2012 έχουν μειωθεί τα φαινόμενα πειρατείας. Μάλλον έχουν ε, εξανεμιστεί σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν πρόκειται για απλά μαγικά αν θέλετε. Έχει να κάνει αυτό με το ότι η συνεργασία ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική. Ομόφωνα επεκτάθηκε η επιχείρηση Αταλάντα για τρία ακόμα χρόνια και αυτό γιατί συντοπίσαμε ότι ε, οι προσπάθειες που είχαμε καταβάλει στο παρελθόν οφείλουν να είναι βιώσιμες. Δηλαδή, αν σταματούσαμε απότομα την Αταλάντα θα είχαμε εκ νέου κάποια φαινόμενα πειρατείας. Γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να συνεχίσουμε την επιχείρηση αυτή η οποία δεν είναι στρατιωτική. Υπάρχει μία συνιστός κατάρτισης του ε, Σομαλικού στρατού στο Μογκαντίσου. αν δούμε όλες αυτές τις διαφορετικές συνιστώσεις, βλέπετε μία ολοκληρωμένη πολιτική για το κέρας Αφρικής, από την οποία ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποια βιώσιμα αποτελέσματα. Όσον αφορά πάντως την πειρατεία, αυτή είχε εξαλειφθεί. Όταν το 2008 ξεκινήσαμε με την επιχείρηση αυτή, είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, 700 ομήρους και πάρα πολλά πλοία που είχαν ε, κατασχεθεί ουσιαστικά, που ήταν ε, σε καθεστώς ομοιρίας. Αν δείτε τα αριθμητικά δεδομένα που έχουμε τώρα, μπορείτε να δείτε πώς έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Και πάλι όμως αυτό δεν είναι τυχαίο οφείλεται στην πολύ επικοδομητική δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όντως βέβαια για την επιχείρηση αυτή τα πράγματα δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν μέσα σε έξι μήνες. Κοιτάξτε, όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, και εκεί έχουμε κάποιες ε, αποστολές. Εδώ ο πολιτικός διάλογος είναι ιδιαίτερα έντονος. Από πλευράς αμυντικού σχεδιασμού δεν μπορούμε να πούμε ότι το Συμβούλιο μας έχει ζητήσει να ξεπεράσουμε τον πολιτικό διάλογο, να προχωρήσουμε δηλαδή σε άλλα επίπεδα. Οι δυνάμεις που έχουμε όμως επιτόπου αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα όσον αφορά τώρα το Σαχέλ, Είμαστε σαφώς πάρα πολύ παρόντες στην περιοχή αυτή, σε καθημερινή βάση επεμβαίνουμε μέσω, για παράδειγμα, της κατάρτισης του στρατού του Μαλή. Στα πλαίσια του ΚΟΠΣ χθες προχθές είπαμε ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και σε μια επέκταση της κατάρτισης αυτής και για την αστυνομία και για το στρατό του Μαλή και υπάρχει μια υποστήριξη και εγχώρια πλέον για τις προσπάθειες αυτές. Τα ίδια ισχύουν και για την Ιγυρία. Έγινε μια αξιολόγηση πρόσφατα της αποστολής αυτής και προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί εκεί για τη Μαυρετανία. Έχουμε πιο συμβατικά κλασικά προγράμματα τα οποία συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Λιβύη τώρα. Προφανώς ε, για τη χώρα αυτή παρακολουθούμε την κατάσταση καθημερινή βάση και διεξάγουμε συνεχείς συζητήσεις και με το ΝΑΤΟ για το πώς μπορούμε να σταθεροποιήσουμε περισσότερο την περιοχή αυτή. Τώρα, θα πρέπει να συζητούμε περισσότερο πριν ή μετά τις αποστολές τις επιχείρησεις αυτές. Όσον αφορά τη Λιβύη έχουμε μια ευρωπαϊκή αποστολή χωρίς τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ επισήμως, παρόλα αυτά συζητήσεις διεξάγονται. Στην Ρώμη, για παράδειγμα, συμμετέχουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ για να προετοιμάσουν την υπουργική διάσκεψη που θα λάβει η χώρα. Όσον αφορά τώρα τις εταιρικέ σχέσεις, ναι, προφανώς έχουμε και εταιρικέ σχέσεις. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα όλους τους εταίρους που έχουν συνεισφέρει στην επιχείρηση αυτή, πάντως ε, η Γεωργία, η Σερβία και πολλές άλλες χώρες ήδη έχουν συνεισφέρει. Δεν τις θυμάμαι τώρα όλες απ' έξω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις να ευχαριστήσουμε τους προσκεκλημένους μας αλλά πριν να κλείσουμε τη συνεδρία να δώσουμε το λόγο στον αντιπρόεδρο της αντιπροσωπείας για τη σχέση με την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ τον κύριο Πάσκο για να μας πει μερικά λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η ανταλλαγή απόψεων που έγινε ήταν αρκετά θετική για τις σχέσεις και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ είναι ένα μόνιμο θέμα στην ημερήσια διάταξή μας. συζητάμε τις σχέσεις αυτές αρκετά συχνά και βεβαίως όποτε γίνεται σχετική συζήτηση ε, ε η, τα θέματα που τίθενται είναι σοβαρά και οι συζητήσεις ενδιαφέρουσες. Τώρα, αυτή η, το Συμβούλιο μας έδωσε κάποιες εντολές ε, σύμφωνα με αυτές πρέπει να ενισχύσουμε την συνεργασία αυτή με το, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και θα πρέπει να δούμε και το σχεδιασμό αν μπορούμε να ευθυγραμμιστούμε τουλάχιστον να συντονιστούμε με τους ΔΕΕ. είδαμε ε, μετά από τη συνεργασία των τελευταίων ετών ότι υπάρχουν <clears throat> και κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιλύσουμε γιατί τα, τα τεχνικά προβλήματα που έχουμε ουσιαστικά επηρεάζουν και τη, τις πολιτικές σχέσεις των δύο οργανισμών. Ε, όπως ελέγχθη, πολλοί πιστεύουν ότι η συνεργασία είναι πολύ πιο σημαντική από τον ανταγωνισμό. Αν δείτε τις δύο από τις τρεις ουσιαστικά δράσεις του ΝΑΤΟ ας πούμε συλλογική άμυνα η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει αναθέτει στο ΝΑΤΟ και αυτό το λέει το άρθρο 42 της συνθήκης της Λισαβόνας ε, ήμουν εισηγητής για μια έκθεση σχετικά, σχετική αυτό είναι γεγονός μετά διαχείριση κρίσεων για το θέμα αυτό μπαίνουμε σε ένα είδος ανταγωνισμό ή άμυλα ίσως θα έλεγα διότι δουλεύουμε στις ίδιες περιοχές και εδώ είναι προφανώς ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ μας. Τώρα ο φίλος μας ο Βανόρντεν όπως και όλοι οι πραγματική Βρετανή ενοχλείται και λέει μα τι στο καλό χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει στρατιωτικές κανότητες δεν έχουμε το ΝΑΤΟ και γιατί το ΝΑΤΟ να μην μπορεί να μας διαθέσει τις ικανότητές του ε, γιατί υπάρχει μια χώρα που λέει όχι τέλος πάντων δεν είναι εδώ ο κύριος τα λέω λίγο στον αέρα όλα αυτά ε, αλλά εδώ θα έλεγα ότι υπάρχει ένα βασικό αμάρτημα από πολύ παλιά. Δηλαδή το ΝΑΤΟ ουσιαστικά τονίζει την συγχαρακτή είναι χαρακτηριστικό για την συνεργασία ε, Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκών χωρών. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έλεγε και ο Σρέμπερ είναι η οικονομικό, οικονομικός ανταγωνισμός αν θέλετε ή ε, ε, η οικονομική πλευρά της όλης, ε, της όλης υπόθεσης Τώρα βέβαια εφόσον έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα ίσως θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε τη σχέση γενικώ το μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης και εμείς βεβαίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αλλιώς βλέπουμε τη σχέση μας με τους Αμερικανούς από ότι οι φίλοι μας της Δυτικής Ευρώπης. Τέλος πάντων για να τελειώνω να πω δύο λόγια για τη Γεωργία. Θα έλεγα ότι στο Βουκουρέστι η Γεωργία χτύπαγε δυνατά την πόρτα του ΝΑΤΟ ε, για να μην την Ουκρανία μαζί για να γίνουν μέλη. Εκεί λοιπόν η Ρωσία έκανε μια επιθετική κίνηση και πήρα ένα κομμάτι αν θέλετε των εδαφών της Γεωργίας για να τα πούμε τα πράγματα όπως έχουν έτσι ε, το ΝΑΤΟ δεν αντέδρασε καθόλου συγχρόνως όμως Ποια είναι η πραγματικότητα τώρα, ότι τώρα η Γεωργία έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να γίνει μέλος κανενός οργανισμού γιατί μέρος του εδάφους της δεν υπόκειται στη κυριαρχία της ε, κυβέρνησης στην Τυφλίδα. Ανοίξει ένα άλλο μπλοκ αν θέλετε. Άντε να βρεις απάντηση σε όλα αυτά. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Και εδώ θα ήθελα να κλείσω να συγχαρώ την υποεπιτροπή, να συγχαρώ τους φίλους μας από τον ΝΑΤΟ που ήρθαν εδώ για να μοιραστούν τις απόψεις τους μαζί μας. Σας ευχαριστώ όλους που αφιερώσατε τόσο χρόνο σε αυτές τις συζητήσεις που κάναμε. Ευχαριστώ πολύ. The meeting is closed. Ευχαριστώ θερμά για τη συνεδρίαση. Something to reassure my colleague. Θα ήθελα να καθησυχάσω το συνάδελφο για κάτι που όλοι ξέρουμε. Αμέσως μετά την επανένωση της Γερμανίας, που έγινε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι όλοι αναμέναμε, για πολλούς μήνες, για να μην πω πολλά χρόνια, είχαμε ρωσικά στρατεύματα στην Ανατολική Γερμανία. Πολύ σημαντική παρατήρηση για μία ακόμη φορά. Μπορούμε να συνεχίσουμε όμως τις συζητήσεις στο διάδρομο.